Λοιπόν, καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Ήδη από χθε ε, σας είχα ανακοινώσει ότι στην Επιτροπή μας έχουμε δύο νέα μέλη, αναπληρωτές, ε, την κυρία Σουτζάνα Μποζάτα και τον κύριο Τζον Στιουαρτ Άγνιου, που είναι παρόντες και οι δύο. Πρόφερα καλά το όνομά σας. Εχθές έκανα και την ε, ανακοίνωση για την παρουσία σας εδώ. Σήμερα σας ε, καλημερίζω και σας εύχομαι καλές εργασίες στην Επιτροπή μας. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε καταρχάς ε, την παρέμβαση του συναδέλφου Γιώζεφ Σάγερ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τη νέα ε, συνταγματική αλλαγή στο Ουγγρικό Σύνταγμα. Ε, να σας πω ότι ήταν πρόεδρος στην ομάδα που ετοίμασε το σχέδιο συντάγματος. Το νέο σύνταγμα ενεκρίθη από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο εχθές. Είχε ζητηθεί η παρουσία και ενό άλλου εμπειρογνώμων από την Ουγγαρία που δυστυχώς δεν είναι μαζί μας. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε καταρχάς τον άδελφο Σάγερ και κατόπιν Εάν ε, η Επιτροπή το θεωρήσει απαραίτητο, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Δεν έχουμε ακόμα βέβαια κείμενο μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες, αλλά πρέπει να γίνει μία πρώτη παρουσίαση, να ακούσουμε και όσοι συμμετείχαν στην Επιτροπή και τον ευχαριστούμε που είναι εδώ να μας δώσει ε, τις ε, ε, πληροφορίες ο ίδιος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω εδώ στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων που είναι νομίζω κατεξοχήν ο χώρος αφού γκράζεστε καινοτομίε και νέα στοιχεία και εξελίξεις στο συνταγματικό δίκαιο υπό την ιδιότητά μου ως πώς το πω, πρώην Προέδρου της ε, Επιτροπής ε, Προετοιμασίας εξ του κόμματός μου, του νέου συντάγματος Ουγγαρίας. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι χθε με μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε το Κοινοβούλιο το νέο σύνταγμα της χώρας που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Πρώτου του 2012. Είναι μεγάλη η συνταγματική προσαρμογή της Ουγγαρίας αυτή. Επί 62 έτη δεν ήταν σε θέση η Ουγγαρία να εγκρίνει νέο σύνταγμα. Το 99 στην αλλαγή ε, έγινε μια βαριά μεταρρύθμιση του συντάγματος για να ε, προσαρμοστεί το σύστημα στις βασικές αρχές κράτους δικαίου και δημοκρατίας. Αλλά Ακόμα, κατά την παραδοχή, κατά την έγκριση μάλλον αυτού του συντάγματος, θεωρήθηκε από την αρχή προσωρινό. Όλα αυτά το 89. Ε, από την αρχή συμμετείχα στην εκπόνηση του συντάγματος και θεωρούσα ότι το νέο εκλεγέν ε, κοινοβούλιο θα ενέκρινε σύντομα νέο σύνταγμα. Δεν έγινε αυτό. 20 χρόνια λοιπόν μετά, η τελευταία από τις κομμουνιστικές, πρώην κομμουνιστικές χώρες, έχουμε πλέον ένα νέο σύνταγμα. Χαίρομαι πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε που δεχτήκατε την πρότασή μου να σας ενημερώσω, όπως είπατε επί του πιεστηρίου για το θέμα αυτό. Θέλω να θυμίσω στους συναδέλφους ότι πριν από αρκετές εβδομάδες στείλαμε το σχέδιο συντάγματος ε, μαζί με την ακρόαση που οργανώσαμε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για ποιο λόγο θέλησα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Γιατί εδώ στην Ευρώπη εμείς είμαστε πολύ στενά συνδεδεμένοι, αλληλένδετοι μεταξύ μας ως χώρες, ε, κοιτάζουμε, παρακολουθούμε πολύ στενά τα συντάγματα μια χώρα της άλλης και ε, αλληλοδιδασκόμεθα. Εμείς ε, στη Ουγγρικό Σύνταγμα εμπνευστήκαμε από τη εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ είχα διατελέσει και μέλος της συντακτικής συνέλευσης και στη συνέχεια παρακολούθησα τα θέματα αυτά από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και τη νομική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνταγματική και προσπαθούμε να ευθυγραμμίσουμε και να εναρμονίσουμε και τη δική μας πρακτική με τα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν λοιπόν κάποια καινοτόμα στοιχεία και ε, είμαι πολύ περήφανος να παρουσιάζω αυτό το σύνταγμα και άλλοι συνάδελφοι μπορεί να χρειαστεί να θελήσουν να ακολουθήσουν το παραδειγμά μας. Ένα στοιχείο που είναι από τα πιο καινοτόμα και τα πιο νεωτερικά, όχι το πρώτο όμως, γιατί ε, στη Γερμανία, στην Πολωνία και στην Ελβετία και σε κάποιες άλλες χώρες ήδη ισχύει. Συνδέεται αυτό λοιπόν με την οικονομική διακυβέρνηση και αντιμετωπίζεται θέματα του χρέους και του δημοσίου ελλείμματος. Είναι η διάρκεια κατάσταση στην Ουγγαρία. Μόλις πριν από λίγους μήνες Ήμασταν σε κατάσταση αντίστοιχη με της Πορτογαλίας τώρα ή και της Ελλάδας πριν από κάποιους μήνες επίσης. Και η Ουγγαρία δεν θα έλεγα ότι είναι η πιο χρεωμένη χώρα στον κόσμο, αλλά είμαστε σε αυτή δυστυχώ την ατυχή ομάδα των πρωταθλητών του χρέους. Δεν είμαστε λοιπόν η πλέον χρεωμένη χώρα, είμαστε χρεωμένοι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από το 2004 ε, είμαστε σε διαδικασία δημοσιονομικού ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπερβολικού ελλείμματος. Αυτό σημαίνει ότι τα τελευταία 20 χρόνια είχαμε ε, κληρονομήσει ήδη από το 90 τεράστιο χρέος κατά την αλλαγή του πολιτεύματος γιατί είχαν συνάψει δάνεια οι κομμουνιστές For Η κυβέρνηση προηγούμενη πολλά χρόνια, δηλαδή είχαμε βαρύ κληρονομιά και βαρύ φορτίο από το παρελθόν. Και αυτό δεν μειώθηκε, αυξάθηκε παρά την ιδιωτικοποίηση και τα άλλα. Ε, λοιπόν, και τα συντάγματα θα πρέπει να αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα όπου είναι πάρα πολύ μείωπες οι πολιτικοί. Τι εννοώ, έχουν ένα ορίζοντα ενός έτους ή δύο ετών ή μέχρι τις επόμενες εκλογές. Ενώ το Σύνταγμα όχι. Και βάλαμε ένα νέο στοιχείο διάκριση των εξουσιών ε, στο Σύνταγμα, ε, στο νέο ε, συνταγματικό δημοσιονομικό συμβούλιο που είναι ένα είδος ελέγχου και παρακολούθησης τύπου checks and balances και σε περίπτωση που δεν συμμορφούνται η κυβέρνηση για τη μείωση του ελλείμματος. Σήμερα το έλλειμμα είναι 82% θα πρέπει λοιπόν να βρούμε νέους τρόπους, ίσως και πειραματισμούς, και να εμπνεύσουμε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που υποφέρουν από τα ίδια προβλήματα. Εδώ κοιτάω γύρω μου, αλλά αυτό μπορεί να αφορά όλους τους συναδέλφους. Κάτι λέει ο κύριος Μέντες Δεβίγκο, δυστυχώς δεν ακούγεται. Ε, έλεγα λοιπόν ότι δεν αρκεί να βάλει κάποιους περιορισμούς ε, των κυβερνήσεων στα συντάγματα και των κρατικών δαπανών για να λυθούν τα προβλήματα του χρέους και άλλα προβλήματα που κληροδοτεί η σημερινή γενιά στις επερχόμενες. Είναι ένα μόνο μέσο και μέτρο και μπορεί να συνδυαστεί με άλλους θεσμούς και με άλλα μέτρα για να αποδώσει. Αυτό πράττει τώρα και ε, η Ουγγρική κυβέρνηση, το νέο Ουγγρικό Σύνταγμα και πολλές χώρες προσπαθούν επίσης να δοκιμάσουν στις δικές τους ε, πρακτικές. Ένα άλλο στοιχείο που είναι επίσης νέο και δείχνει ότι το Σύνταγμα είναι Σύνταγμα του 21ου αιώνα ήδη έχει ενσωματώσει πολλά στοιχεία της συνθήκης της Σαβώνας. Η αναφορά στην Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μία, βρύφη αναφορών και δεν είναι μόνο τυπική. Ήδη από το προήμιο παραπέμπουμε ε, στις ε, ευρωπαϊκές αξίες και αρχές. Αλλά ε, στο συνταγματικό κείμενο αυτό καθ' αυτό λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αναφέρουμε ως το πλαίσιο της ανάπτυξης της χώρας μας στο μέλλον. Είναι και σημείο αναφοράς. Και βέβαια ορίζουμε πώς εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο στην Ουγγαρία, τι γίνεται με τις ε, τοπικές περιφερειακές εκλογές και πώς μπορούν να συμμετέχουν στη συνταγματική ζωή της χώρας οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλη λοιπόν αναφορά και σημαντικό πλαίσιο ανάπτυξης ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επόμενο σημείο Um, uh, Hungary is proud of is... Uh, ένα άλλο στοιχείο που είμαι και εγώ προσωπικά περήφανος αλλά και η Ουγγαρία ολόκληρη είναι η αρχή της βιωσιμότητας και εφορίας. Of... Τρεις είναι οι αρχές εδώ εφορίας που βεβαίως είναι ένα νέο στοιχείο και μια νέα έννοια του 21ου αιώνα. Η βιωσιμότητα του προϋπολογισμού, το είπα ήδη αυτό, σημαντική κατευθυντήρια ε, γραμμή δεν το ορίζουμε απλώς ως γενική αρχή στον προπολογισμό, αλλά ε, δημιουργούνται και θεσμοί για να υποστηρίξουν αυτή τη συνταγματική αρχή και το κείμενο του συντάγματος. Για πρώτη φορά, όπως σα είπα, και είναι καινοφανέ αυτό, ε, αναφέρεται η διάκριση των ε, εξουσιών και ένα σύστημα ελέγχων και αντιβάρων. Βαρών, το θέμα δεν είναι ίσως κερδισμένο ο προπολογισμό. Αυτό είναι γενική αρχή. Οι πάντε οφείλουν. Αλλά ε, εισάγουμε και το στοιχείο τη ευθύνη για τις επόμενες γενιές. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να εφαρμόζεται ω γενική αρχή. Η αηφορία της δημοκρατίας της χώρα μας, αλλά και ευρύτερα. Επίσης, αυτό μπορεί να ενδιαφέρει και την Επιτροπή μας εδώ για συζήτηση ε, περαιτέρω. Δεν θέλω εγώ να τη σταματήσω. Είναι το πώς μπορούν οι γονείς να αποφαίνονται και να μιλούν στο όνομα των παιδιών τους. Αυτό δεν το βάλαμε στο Σύνταγμα, όπως γράφει ο Guardian ή άλλες εφημερίδες. Ήταν στο προσχέδιο, αλλά ε, έγινε ευρεία διαβούλευση με ερωτηματολόγιο 12 ερωτήσεων που σε κάθε ουγγρικό νοικοκυριό και απάντησαν περίπου ένα εκατομμύριο Ουγγροί. Ήταν ανώνυμο δε το ερωτηματολόγιο. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω δημοσκόπηση γιατί δεν είναι δείγμα. Το στείλαμε σε όλους και όσοι ενδιαφέρονται έστειλαν και απάντηση. Αλλά μόλις 25% των ε, ε, όσων απάντησαν υποστήριξαν αυτό. Κοιτάξτε, είναι από τα αγαπημένα μου θέματα και θα ήθελα να γίνει και ακρόαση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλοί θεωρούν και στην Ουγγαρία όταν το άκουσαν για πρώτη φορά ότι το λέμε για αστεία, ότι είναι ανέκδοτο. Καθόλου ανέκδοτο δεν είναι. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον νόμο, με την εκπαίδευση. Δεν λέω ότι πρέπει να το συζητήσουμε τώρα. Uh, ε, σε λίγους μήνες ε, μπορώ να το ξαναφέρω προς συζήτηση, ιδιαίτερα και σε ό,τι αφορά τη δημογραφική βιωσιμότητα και εφορία. Και Επίσης το συνταγματικό ε, κείμενο αυτό δεσμεύεται να υποστηρίζει και να βοηθάει οικογένειες και πολίτες με παιδιά ε, ο ορισμός ε, του γάμου και ο ορισμός της οικογένειας δεν είναι κάτι που ορίζει το Σύνταγμα γιατί ακούσαμε και τέτοιες κατηγορίες και αιτιάσεις πρόσφατα και το είδαμε και στις εφημερίδες ότι ε, εξαιρούνται οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι εναλλακτικέ μορφές οικογένειας. Καθόλου δεν το αναγράφει αυτό το γράμμα του Συντάγματος. Είναι παρερμηνίες ένα άλλο θέμα που θα σας ενδιαφέρει, γιατί το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα εδώ στο Κοινοβούλιο, είναι θέμα περιβάλλοντος. Η αηφορία από πλευράς περιβάλλοντος. Είναι πολλές οι αρχές που εφαρμόζουμε και ε, τα βασικά επιτεύγματα είναι μεταξύ άλλων η αρχή του «Ο πληρώνει» Ο περιορισμός ε, εναπόθεσης ε, ε, τοξικών και άλλων αποβλήτων στην επικράτεια της χώρας, υποστήριξη της βιοπικιλότητας. Πρέπει να σας πω ότι κατατέθηκε και μια τροπολογία στο Σύνταγμα που περιορίζει ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Η χώρα είναι ελεύθερη ε, μεταλλαγμένων και το γράψαμε και στο Σύνταγμα για να κατοχυρωθεί. Θα σταματήσω εδώ, Πρόεδρε, γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι πολλές ερωτήσεις και με χαρά να σας απαντήσω από πρώτο χέρι, γιατί στην όλη διαδικασία που διήρκησε 10 μήνες ήταν μεγάλη παραπληροφόρηση, παραπλανήσεις ή παρερμηνίες ε, και για να είναι σωστά ενημερωμένο το ευρωπαϊκό κοινό ε, θα πρέπει να ενημερωθούμε σωστά. Όχι εδώ σε αυτή την ομίγυρη, αλλά ε, κάποιοι δημοσιογράφοι που γράφουν τέτοια άρθρα δεν γνωρίζουν ούτε τις ίδιες τους τις χώρες το Σύνταγμα και γράφουν για το Ουγγρικό. Τώρα δεν χρειάζεται να γίνει καμιά μελέτη ή συζήτηση. Βέβαια, Κάθε σύνταγμα είναι υπόθεση της κυριαρχίας ενός κράτους. Αλλά μπορούμε να συζητήσουμε τις γενικές και κοινές αρχές. Κάτι άλλο. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό και παρακάθεται εδώ ο ίνικομέντες Μέντες Δεβίγκο που ήταν από τους συντάκτες του Χάρτη Θεμελιωδών Ελευθεριών. Ε, ε, Χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λοιπόν στην Ουγγαρία βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη και είναι το πιο σύγχρονο κείμενο του 21ου αιώνα. Και ακολουθούμε. Βέβαια όχι κατά γράμμα, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη παράδοση αποφάσεων συνταγματικού δικαστηρίου ε, και πολύ ε, πλούσια εμπειρία την τελευταία 20 ετία. Η προστασία της ιδιοκτησίας και τα λοιπά είναι πράγματα που απορρέουν από τη συνταγματική μας εμπειρία, από το συνταγματικό δικαστήριο. Είναι μεγάλη λοιπόν υπόθεση και μεγάλο επίτευγμα μετά από 22 χρόνια να μιλάει ε, για τα δικαιώματα του πολίτη το Σύνταγμα πρώτο. Ο Λόγκλι ή το 49 ο δικτάτοράς μας που ενέκρινε τότε το σταλινικό σύνταγμα πρώτα το κόμμα, μετά το κράτος και τελευταίος ο πολίτης κάποια στιγμή. Και δυστυχώς το 1989 όταν ε, αλλάξαμε το σύνταγμα και εγώ συμμετείχα εκεί στην αναθεώρηση δεν είχαμε ούτε το χρόνο ε, ε, ούτε τη δυνατότητα να αλλάξουμε ολόκληρη τη δομή του συντάγματος οπότε είχε μείνει στο τέλος ο πολίτης. Λοιπόν, φιλοσοφικά είναι μεγάλη ανατροπή αυτό. Το Σύνταγμά μας βασίζεται πρώτα στα δικαιώματα του πολίτη και όχι στο πανίσχυρο και παντοδύναμο κράτος. Ευχαριστώ που μου δώσατε, Πρόεδρε, λοιπόν, την ευκαιρία να σας ενημερώσω για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να κάνουν τα σχόλιά τους και να μας βοηθήσουν για την επόμενη φάση του Ουγγρικού Συντάγματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζάγερ για την ε, πλήρη αυτή παρουσίαση. Νομίζω ότι καθήκον μου είναι καταρχάς να οργανώσω λίγο τη συζήτηση, διότι θα ήθελα να την ολοκληρώσουμε στις 10 για να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να ακούσουμε τις επικεφαλείς των διαφόρων πολιτικών ομάδων και εάν υπάρχει χρόνος να ακούσουμε και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Ο κύριος Γκερέρο έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Σάγερ, ο οποίος ε, ήρθε εδώ στην Επιτροπή μας σήμερα. Να επισημάνω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, γι' αυτό θα πρέπει να οργανώσουμε και νέες συζητήσεις για το Ουγγρικό Σύνταγμα. Αυτή τη στιγμή θα διαθέτουμε και το κείμενο μεταφρασμένο σε διάφορες γλώσσες. Θα ήθελα να επισημάνω καταρχάς ότι όλα όσα θα πω στην παρέμβασή μου απορρέουν από το γεγονός ότι αναγνωρίζω το ε, γεγονός ότι ο Ουγγρικός λαός είναι κυρίαρχος και μπορεί να οργανωθεί όπως θεωρεί απαραίτητο και το γεγονός ότι ο κυρίαρχος αυτός λαός, ε, ο λαός αυτός είναι κυρίαρχος, θα πρέπει να καθορίζεται εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει λοιπόν να τηρούνται οι αρχές, οι αξίες και οι δυνατότητες ε, της κοινή οργάνωσης που, στην οποία ανήκουμε όλοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα καταρχάς να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για την ε, συνταγματική διαδικασία της Ουγγαρίας, συγκρίνοντάς την με τη συνταγματική διαδικασία στην ε, Ισπανία μετά από τη λήξη της δικτατορίας του Φράνκο και κατά τη μετάβαση στη δημοκρατία. Η Ισπανία από τις αρχές του 19ου αιώνα είχε 7 διαφορετικά συντάγματα. Κάποιοι εξ αυτών ε, ψηφίστηκαν και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Ζήσαμε ο, ολοκληρωτικά καθεστώκα και κανένα από αυτά τα συντάγματα δεν έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία του ε, ισπανικού λαού. Κάποια ήταν καλύτερα και κάποια χειρότερα, αλλά έλειπε το πιο σημαντικό στοιχείο, η κοινωνική συνένεση. Κάθε φορά δινόταν η ερμηνεία του συντάγματος ενός κόμματο και το απέριπτε η άλλη πλευρά της κοινωνίας που θεωρούσε ότι δεν ε, το εκπροσωπούσε αυτό το σύνταγμα. Στις εκλογέ του 1978, που ήταν οι πρώτε δημοκρατικέ εκλογέ. Ε, είχαμε μια συντακτική συνέλευση που αποτελούνταν από 7 μέλη, 4 εκ των οποίων ήταν από κόμματα της αντιπολίτευσης. 4 από τα 7 μέλη. Η συζήτηση λοιπόν για το Σύνταγμα ολοκληρώθηκε με ψηφοφορία υπέρ του Συντάγματος και είχαμε 92% ψήφων και 96% στο, στο Κοινοβούλιο στην Ισπανία και υπήρξε και ευρύτατη υποστήριξη στο δημοψήφισμα που έγινε στην Ισπανία. Και αυτό το σύνταγμα είναι γνωστό στην Ισπανία ως το σύνταγμα της συνένεσης. Με αυτό το σύνταγμα κυβέρνησαν στη συνέχεια τρία διαφορετικά πολιτικά κόμματα στην Ισπανία και κάποιοι εξ αυτών όπως το Σοσιαλιστικό Κόμμα κυβέρνησε, εκχώρησε την εξουσία και ήρθε στα πράγματα. Αυτή τη στιγμή το Σύνταγμα είναι πιο ισχυρό από ποτέ. Πρόκειται για το Σύνταγμα το οποίο έχει τη μεγαλύτερη ε, διάρκεια στη συνταγματική ιστορία της Ισπανίας. Έχει προκύψει από ευρεία πολιτική συνένεση και από ευρεία αδημαϊκή συνένεση. Και είναι ένα σύνταγμα το οποίο περιλαμβάνει όλους. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω μία σύγκριση με την όλη διαδικασία στην Ουγγαρία. Ήταν απαραίτητο αυτό το σύνταγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, θα πρέπει να το απαντήσουν οι Ούγγροι και δεν θα πω εγώ την άποψή μου. Αυτό που ξέρω είναι ότι σίγουρα στην Ουγγαρία υπάρχει διχογνωμία για το κατά πόσον είναι απαραίτητο ή όχι αυτό το νέο σύνταγμα. Υπάρχει ένα σκέλος το οποίο θεωρεί ότι το σύνταγμα αυτά ε, υπενθυμίζει αυτό του 1949 και υπάρχει και ένα σκέλος το οποίο θεωρεί ότι αυτό το Σύνταγμα δεν ήταν τόσο απαραίτητο δεδομένου ότι έγιναν πολλές μεταρρυθμίσεις το 1989 ε, όταν ε, έπαψε να υπάρχει ο κομμουνισμός στην Ουγγάρια. Δεν θα πω περισσότερα γιατί οι Ούγγροι είναι αυτοί οι οποίοι θα πούν κατά πόσο απαιτείται ή όχι ένα νέο σύνταγμα. Αυτό το οποίο βέβαια είναι διαμφισβήτητο είναι ότι ήταν ε, κομματική ε, υποστήριξη. Δεν υπήρχε ε, μία συντακτική συνέλευση, μία ομάδα η οποία εκπώνησε υποστηριξη δεν υπηρχε μια συντακτικη συνελευση σύνταγμα και να συμπεριλάμβανε μέλη άλλων κομμάτων. Συμμετείχε μόνο το κυβερνόν κόμμα. Το κυβερνών κόμμα ουσιαστικά είναι το μόνο κόμμα το οποίο υπερψήφισε το Σύνταγμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων ε, στην Ουγγαρία και είναι γνωστό ότι οι Ούγγροι πολίτες δεν μπόρεσαν να εκφράσουν την άποψή τους ε, για το Σύνταγμα αυτό μέσω δημοψηφίσματος όπως γίνεται συνήθως όταν έχουμε συνταγματική μεταρρύθμιση. Το κυβερνών κόμμα βέβαια μπορεί να πει ότι έχει πλειοψηφία και μπορεί να υπερψηφίσει το Σύνταγμα και αυτή η πλειοψηφία νομιμοποιείται διότι πρόκειται για τη λαϊκή βούληση. Θα πρέπει όμως να πω ότι αυτό το οποίο συνήθως ισχύει και θα έπρεπε να ισχύει για τα ε, κυβερνητικά προγράμματα, δεν θα πρέπει να ισχύει και για τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Το Σύνταγμα θα πρέπει να ε, αντικατοπτρίζει τις απόψεις της πλειοψηφίας της κοινωνίας και θα πρέπει να μπορεί να υπάρχει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει ο καθένας να εκφράσει το πολιτικό του πρόγραμμα. Και δεν θα πρέπει κάποιος να εκμεταλλευτεί μια ισχυρή αλλά μεταβατική πλειοψηφία για να παγώσει ένα ε, πολιτικό σύστημα το οποίο πολύ δύσκολα μπορεί να τροποποιηθεί. Η ιστορία αποδεικνύει ότι όταν δεν συμπεριλαμβάνει τους πάντες σε αυτό το πλαίσιο, οδηγούμαστε στην αστάθεια και στις συγκρούσεις εντός της κοινωνίας. Η άποψή μου λοιπόν για τις συγκεκριμένες πτυχές ε, του συντάγματος θα διατυπωθεί, αν υπάρχει δυνατότητα, όταν θα γνωρίζουμε επακριβώς τι περιλαμβάνει το Σύνταγμα της Ουγγαρίας. Αλλά νομίζω ότι είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η διαδικασία είναι η διαδικασία που θα αναμενόταν από μια χώρα που ανήκει, όπως είπα, στο συνταγματικό μας πλαίσιο και εστερνίζεται τις αξίες που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει πολιτική πλειοψηφία και νομιμότητα, σαφώς. Υπάρχει νομιμότητα για να εγκρίνουμε το Σύνταγμα, σαφώς. Αλλά νομιμότητα για το κατά πόσον περιλαμβάνει το μέγιστο της κοινωνίας υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσον υπάρχει και το τι θα γίνει στο μέλλον με διαφορετικές κυβερνήσεις και διαφορετικά πολιτικά προγράμματα είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα πρέπει να ξαναδούμε διότι εάν το Σύνταγμα θα πρέπει να δούμε αν το σύνταγμα το οποίο εγκρίθηκε χθε από την Ουγγαρία ε, εκπροσωπεί όλους και όχι μόνο την πλειοψηφία που βρίσκεται στο κυβερνών κόμμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γκερέρο. Στη συνέχεια ζητήσει το λόγο ο κύριος Νταφ. Κύριε Πρόεδρε. Αντίθετα μετά όσα είπε ο ο κύριος Γκερέρο, η χώρα που γνωρίζω εγώ καλύτερα δεν έχει καμία απολύτως εμπειρία από τη σύνταξη συνταγμάτων. Επομένως θα πρέπει να πω ότι ζηλεύω ιδιαίτερα τον κύριο Σάγερ, ο οποίος είχε την ευκαιρία αυτή να καταφέρει να πετύχει κάτι τόσο σημαντικό. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο βέβαια ότι στην δική μας την Επιτροπή η ανησυχία μας έχει δύο πτυχές. Πρώτον, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ότι ε, η σχέση ανάμεσα στην Εθνική Σταγματική Μεταρρύθμιση και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ε, μεταρρύθμιση της, ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όντως υφίσταται, ότι συνάδουν αυτά τα δύο. και ότι ε, τα μεταρρυθμιστικά μέτρα τα οποία προβλέπονται τόσο στη συνθήκη όσο και στο εθνικό σύνταγμα ή τα εθνικά συντάγματα δεν θα οδηγήσουν σε μη αναγκαίες ε, συγκρούσεις, αντιθέσεις ή αντιφάσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι ε, οποιαδήποτε εθνική μεταρρύθμιση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις που υπάρχουν με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Ως προς αυτό λοιπόν θα ήθελα να μου δώσει ο κύριος Σάγερ κάποιες εξηγήσεις για τη ρήτρα εκείνη στο Σύνταγμα, η οποία φαίνεται να αναφέρεται στην Ουγγρική Διασπορά, να υποστηρίζει, να προωθεί τη Διασπορά αυτή. Τη ρήτρα αυτή, η οποία προωθεί ουσιαστικά την εθνική ταυτότητα των ατόμων εκείνων που είναι Ουγγρικής καταγωγής, αλλά ζουν διαμένουν εκτός των συνόρων της ε, Ουγγρικής Δημοκρατίας. Νομίζω ότι ε, υπάρχουν σαφώς κάποια σημεία στο Σύνταγμα αυτό τα οποία μπορούμε να χαιρετήσουμε και να αποδεκτούμε. Ε, στο πλαίσιο βέβαια της κατανοησής μας αυτή τη στιγμή του σχεδίου συντάγματος ή μάλλον αν θέλετε το κειμένου που εγκρίθηκε χθες, το γεγονός ότι υπάρχει μια ρήτρα που αναφέρεται στη συμβολή της Ουγγαρίας όσον αφορά το στόχο της ενότητας, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ρήτρα. Σε καμία περίπτωση δεν θα βλέπατε κάτι ανάλογο σε ένα Βρετανικό σύνταγμα. Επίσης, το γεγονός ότι απαγορεύονται τα δημοψηφίσματα και ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικύρωση τροποποιήσεων στις ευρωπαϊκές συνθήκες, στις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διάταξη αυτή, η ρήτρα αυτή μου φαίνεται ότι είναι επικοδομητική και ουσιαστικά συνάδει πλήρως με τις υποχρεώσεις της ε, εν λόγω χώρας ως προς το σεβασμό της συνθήκης. Επίσης, η αναφορά που έγινε ε, στο χάρτη είναι πολύ σημαντική, αλλά βέβαια η συμπερίληψη είναι μόνο μερική. Και καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιες συγκρούσεις με το Σταγματικό Δικαστήριο στη Βουδαπέστη και με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. και νομίζω ότι προβλέπεται λογικά από τους συντάκτες του συντάγματος ότι η απουσία αναφορά στον σεξουαλικό προσανατολισμό και η ε, απουσία αναφορά στην κατάργηση της θανατικής ποινής, αυτά τα δύο ζητήματα μπορούν να προκαλέσουν ε, προβλήματα. Επίσης, η πρόταση να μπορούν να ψηφίζουν ε, οι μητέρες εξ ονόματος των παιδιών τους είναι μια πρόταση που κατά την άποψή μου βάλει κατά της πράξης άμεσων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της πράξης του 1976. Αν τελικά εφαρμοστεί για τις ευρωπαϊκές εκλογές η διάταξη αυτή και νομίζω ότι υπάρχει και μια ρήτρα που λέει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αυτός που θα καθορίσει την ημερομηνία για τη διεξαγωγή των ευρωπαϊκών εκλογών. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν συμμορφώνεται με την κοινοτική νομοθεσία. Όσον αφορά τώρα την, τις διατάξεις που έχουν να κάνουν με την δημοσιονομική πειθαρχία, τι να σας πω, καλή τύχη. Καλώ, ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Χέφνη. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σας κύριε Σάιερ για την εισαγωγή σας. Σωστό το θεωρώ και απαραίτητο πολύ περισσότερο. Εμείς ως Συνταγματική Επιτροπή του Κοινοβουλίου να ασχολούμαστε με τα συντάγματα των κρατών μελών μας, όπου έχουμε νέες εξελίξεις και θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό εδώ το εξής ερώτημα. τα συντάγματα στην Ευρώπη συγκλίνουν ή αποκλίνουν μεταξύ τους, ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη δημοκρατία, τη διάκριση των εξουσιών, ε, το κράτος δικαίου, το checks and balances, αυτό που είπατε, τους ελέγχους και την ε, παρακολούθηση εξουσίας και πολύ γρήγορα μάλιστα έρχεστε, μόλις εχθές εγκρίθηκε το Σύνταγμα και μπορούμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συζητούμε ήδη. Με προσοχή άκουσα τα όσα είπατε και έχω μερικές πολύ μεγάλες επιφυλάξεις όσο και ανησυχίες που θα ήθελα να σας αναφέρω για να σας υποβάλω ε, υποτύπων ερωτήματος. Ένα στοιχείο που για μένα είναι το σημαντικότερο όλων. Οι κυβερνήσεις εκλέγονται για μια θητεία, για ένα χρονικό διάστημα από το λαό για να κυβερνούν τη χώρα σωστά. Στη συνταγματική θεωρία γίνεται η διάκριση ε, ανάμεσα ε, στη συντακτική εξουσία και στην συντεταγμένη εξουσία. Για τον τρόπο με τον οποίο εκλέγεται λοιπόν συντακτική εξουσία στη δημοκρατία, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι ο λαός. Και το να δημιουργείται ένα σύνταγμα δεν θα πρέπει να διέπεται από τον καιροσκοπισμό, τον οπορτουνισμό ενός κόμματος ή μιας πολιτικής παράταξης. Αλλά πάντα όλες οι πολιτικές δυνάμεις να μπορούν να συμμετέχουν. Και ε, αυτό ε, είναι και διαχρονικό και δημιουργεί ένα πλαίσιο συντάγματος το οποίο μπορεί να ακολουθεί μια κυβέρνηση δεξιά, αριστερή, κεντρώα κτλ. Όχι για εκάστοτε κυβέρνηση ε, κατά το δοκού να φτιάχνει ένα σύνταγμα. Ε, αλλά να υπάρχει συνένεση στον πληθυσμό να υπερβαίνει κατά πολύ το στενό πλαίσιο της κομματικής παράταξης της κυβέρνησης και να το ασθενίζεται όλος ο λαός. Βέβαια αυτό είναι και η τέχνη ε, των ε, ε, κυβερνώντων να κάνουν με τέτοιο τρόπο τις συζητήσει και τις διαδικασίες ώστε να συμμετέχουν όλοι και να αντιλαμβάνονται όλοι και να αισθάνονται ότι και τα συμφέροντά τους και τα ενδιαφέροντά τους και οι απόψεις τους λαμβάνονται υπόψη. Έχω μεγάλες επιφυλάξεις και ανησυχίες εάν έγινε αυτό και κατά πόσο στην ε, Ουγγαρία και αν υπήρχε καν η βούληση να γίνει. Αυτό το στοιχείο του ερωτηματολογίου για μένα μπορεί να είναι καινούριο και ενδιαφέρον, αλλά και ιδιαίτερα προβληματικό. Αν κοιτάξετε τις ερωτήσεις, που στέλνετε με επιστολή στους πολίτες. Ας πούμε, ρωτάτε τους πολίτες, είστε υπέρ ή κατά του συντάγματος που γράφουν κάποιο, το γράφουν κάποιοι πολιτικοί. Αυτό δεν το ρωτάτε χρησιμοποιείτε τους πολίτες ως μαντίο παρά ως κυρίαρχο λαό που θα πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο ως συντακτική εξουσία. Ο λαός καθορίζει το Σύνταγμα, από το λαό απορρέει το Σύνταγμα. Να σας πω τώρα τα σημεία που με ανησυχούν πιο πολύ. Ich habe vorhin gesagt, Sie haben von... Προηγουμένως είπατε ότι ο λαός σας έδωσε πολύ ε, εμπιστοσύνη. Για τέσσερα χρόνια όμως, για να υγείστε της χώρας. Έχω την τάση να πιστεύω ότι αυτή την εξουσία που σας έδωσε ο λαός, η κυβέρνησή σας θέλει να την επεκτείνει και χρονικά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Με συνταγματική ρύθμιση μειώνεται τη θητεία των δικαστών και των εισαγγελέων αυτό δημιουργεί μεγάλες ε, αμφιβολίες και επιφυλάξεις για τη δικαστική εξουσία, για τη διάκριση των εξουσιών. Μα η, δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη από την εκτελεστική και την νομοθετική. Επίσης μιλήσατε για τις μεγάλες προσπάθειες που κάνετε να μειώσετε το έλλειμμα του προπολογισμού. Τα κριτήρια του Μαστρίχτ λέτε θέλετε να τα τηρήσετε στο μέλλον. Και στο τέλος είπατε ότι έχετε πείγνωση ότι σημασία δεν έχει το τι λέει το Σύνταγμα, αλλά τι θα συμβεί επί τη ουσία. Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν προβλήματα ε, δημοσιονομικά, τείνουν να αυξήσουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Και στην Ουγγαρία το αυξάνεται κατά 8 έτη όχι για όλο τον πληθυσμό που θα ξεσηκωνότανε, αλλά για ένα κλάδο επαγγελματικό που είναι οι δικαστές και οι ε, εισαγγελείς. Και επίση κάποιοι άλλοι απολύονται και προσλαμβάνεται άλλους, ικανοί άνθρωποι κατά τα άλλα, δεν λέω. Αλλά δημιουργείται η εντύπωση ή η υποψία ότι διορίζεται κάποιος που είναι ευνοϊκά διακείμενοι απέναντί σας. Για ποιο λόγο να ορίζει το Σύνταγμα ποια θα είναι η θητεία των δικαστών και των εισαγγελέων και μόλις αλλάξει ο χρόνος συνολικά να σαρώσουν οι αλλαγές στην ηγεσία και στη δικαιοσύνη την ίδια. Και έχετε περιορίσει πάρα πολύ και όχι μόνο τη θητεία των δικαστών και των εισαγγελέων, αλλά και τις δικαστικές εξουσίες. Έχετε τα δύο τρίτα της Βουλής και ε, παίρνετε αποφάσεις και ο κόσμος πιστεύει ότι θέλετε να βάλετε δικούς σας δικαστές και για να μιλήσω λίγο και για το ποδόσφαιρο. Η Γερμανία και η Ουγγαρία έχουν κοινή ποδοσφαιρική ιστορία και ενδιαφέρουσα. Εγώ πιστεύω ότι οι πολίτε ψηφίζουν πολιτικού για να είναι ομάδα και να λειτουργούν ομαδικά στο γήπεδο. Για να παίξει όμω ω ομάδα θα πρέπει να έχει συμφωνήσει από κοινού του κανόνε. Και ποιο φροντίζει να ελέγχει τους κανόνες. Και εγώ αρχίζω και φοβάμαι και ανησυχώ όταν μια ομάδα που είναι πολύ επιτυχή στο γήπεδο Ξαφνικά αποφασίσει λοιπόν να αλλάζουμε του κανόνε και αλλάζουμε και το διαιτητή. Στο μέλλον θα λέμε εμεί ποιο θα είναι ο διαιτητής και δεν δεχόμαστε διαιτητές που να έχουν ορίσει άλλοι. Αυτό στην κοινή Ευρώπη από πλευρά κράτου δικαίου διάκριση των εξουσιών να ενισχύει βαθύτατα. Το είπατε και εσείς ο ίδιος ότι θέλετε να ενισχύσετε τον έλεγχο και την εξισορρόπηση. αυτό το balance το έχετε χάσει και το checks έχετε χάσει γιατί έχετε μειώσει ε, την ε, βούληση του κυρίαρχου λαού, έχετε αποκλείσει δημοψηφίσματα, δεν ξέρω μήπως μπορείτε να μας τα εξηγήσετε. Ελπίζω να διασκεδάσετε τις ανησυχίες και τους φόβους μου και να είναι αβάσιμοι, πάντως ανησυχώ. Θα πρέπει να αρχίσω να σας συστήνω να είστε λίγο πιο λακωνικοί. Ο κύριος Σόλτς. Ähm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους συναδέλφους μου. Και βέβαια είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και λεπτή συζήτηση σχέση ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου και πολιτική κυριαρχία και ανεξαρτησία της κάθε χώρας, έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν πρόκειται για τόσο σημαντικά θέματα όπως είναι ε, ένα σύνταγμα, η ψήφιση ενός συντάγματος. Βεβαίω καλό είναι και σωστά υπόθηκε ότι πρέπει να συζητούμε και εμεί στην Επιτροπή μας για τα τεκτενόμενα τα κράτη-μέλη, γιατί έχουν και επίδραση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο κοινοτικό δίκαιο. Για το λόγο αυτό, ε, τρία σύντομα σχόλια. Το Σαββατοκύριακο ήμουν στη Βουδαπέστη σε μια διάσκεψη ε, Ρωμά και εκεί εκφράστηκε μεγάλη ανησυχία για τη μελλοντική πολιτική και ε, νομοθετική κατάσταση στη χώρα. Εξού και το ερώτημα. Όταν λέμε ότι οι πολίτες χάνουν την εμπιστοσύνη τους ε, στην πολιτική και την απαξιώνουν, και το λέμε συχνά και στην Ευρώπη. Αν η πολιτική λοιπόν δεν φροντίζει να είναι διαφανής ο τρόπος με τον οποίο παίρνει τις αποφάσεις τους, εάν οι πολίτες αισθάνονται αποκλεισμένοι, αυξάνεται το χάσμα που μας χωρίζει από τους πολίτες. Και αυτό ε, ισχύει κατεξοχήν στην ψήφιση ενός συντάγματος. Το είπαν και πολλοί συνάδελφοι προηγουμένως. Και θα με διέφερε εμένα. Γιατί έχοντας και την εμπειρία του ναυαγίου ε, του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, της Συνταγματικής Συνθήκης, γιατί ε, δεν επιλέξατε ανοιχτά το δρόμο του δημοψηφίσματος για το νέο σύνταγμα στην Ουγγαρία. Έτσι ώστε ο λαός που είναι κυρίαρχος, ο λαός είναι ο κυρίαρχος, το ακούσαμε μόλις, να έχει λόγο για το σύνταγμα και άμεσα για το μελλοντικό του σύνταγμα να συναποφασίζει. Και αυτή η λαϊκή βούληση για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική και το λέω και συνειδητά. Διότι προέρχομαι από ένα τμήμα της Γερμανίας που το 1989 αποφάσιζε μόνο του το κόμμα να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά τέτοια διαίρεση. Αυτό που είχε πει η Ρόζα Λούξεμπουργκ, ότι η ελευθερία σημαίνει πάντα και την ελευθερία εκείνου που σκέφτεται διαφορετικά από μένα. Αυτό δεν θα πρέπει να ισχύει και για το σύνταγμα ενός κράτους. Το λέω ξεκάθαρα και ειλικρινά. Θα ήταν πολύ σημαντικό για μένα να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για όλους τους πολίτες. Κάθε ε, άντρα και κάθε γυναίκα που είναι πολίτης της Ουγγαρίας. Στη συνέχεια. Στο βαθμό που μπόρεσα να παρακολουθήσω το κείμενο με την προσωρινή μετάφραση, μερικά βασικά κοινωνικά δικαιώματα που ήταν κατοχυρωμένα στο Σύνταγμα έχουν εξαφανιστεί. Παράδειγμα, το ρητό δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, τη δημιουργία συνδικάτων, των απεργιών. Τα βασικά στοιχεία, ελευθερία του συνέρχεστε, δεν αναφέρονται τόσο ρητά ως κοινωνικά δικαιώματα στο Σύνταγμα. Άλλο θέμα. Εάν δούμε τα σημεία επαφής ε, της Εθνικής Συνταγματικής Μεταρρύθμισης με την ε, μεταρρύθμιση των συνθήκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να πούμε ότι η Ουγγαρία Βάσει του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να συνεισφέρει στη μετεξέλιξη και στη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό έχει να κάνει και με τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Κάθε είδους και χρειάς. Ε, μέχρι και το ε, σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά και όχι μόνο. Και τα δικαιώματα των εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων με την ευρύτερη έννοια. Θα πρέπει να έχουν την ελευθερία των δικαιωμάτων τους. Και επίσης τι είναι αυτό που λέτε για την εκπροσώπηση Ούγγρων που ζουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πώς θα συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Καλώς. Ο λόγος τώρα στον κύριο Μέντες Τεβίκο. Ευχαριστώ. Θες να μιλήσεις πριν από μένα. Πρώτα ο Έλμαρ. Πάντα ο Έλμαρ προηγείται. Hoffentlich werde ich so alt Hoffentlich. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ λοιπόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σάγερ για την ε, ταχύτατη παρέμβασή του. Νομίζω ότι ούτε 24 ώρες δεν πέρασαν πριν από την έγκριση του συντάγματος και είναι ήδη εδώ και μας μιλά για το σύνταγμα. Νομίζω ότι πρόκειται λοιπόν για καλή πρωτοβουλία. Αναγνωρίζω βέβαια ότι δεν γνωρίζω τι λεπτομέρειε του κειμένου, ούτε καν τα πιο γενικά. Φαίνεται ότι άλλοι συνάδελφοι έχουν ήδη το κείμενο αναχείρας, εγώ αναγνωρίζω ότι δεν το διαθέτω. Θα κάνω λοιπόν πολύ γενικέ παρατηρήσει. Καταρχά να πω ότι θεωρώ καλό ότι γίνεται η συζήτηση αυτή εδώ με πρωτοβουλία του κυρίου Σάγκερ γιατί καταδεικνύει ότι υπάρχει διάθεση να εξηγήσει, να μιλήσει, να μα αιτιολογήσει πράγματα. Δεύτερον, εγώ θεωρώ ότι τα συντάγματα, και ακούστηκε εδώ, δεν θα πρέπει να είναι σύνταγμα της κυβέρνησης, ε, του κόμματος που έχει την κυβέρνηση, γιατί δεν είναι και μακρόβια τα πολιτικά κόμματα. Ξέρετε ότι συνήθω οι πλειοψηφίε αλλάζουν και εάν το σύνταγμα αυτό είναι το σύνταγμα ενός κόμματος και όχι του λαού, τότε θα έρθει το επόμενο κόμμα και θα το αλλάξει και αν όντως ισχύει αυτό δεν είναι καλό σίγουρα, είναι κακό. Δεν θα πρέπει όμως να είμαστε υπερόπτες ε, προς τους υπολείπους, ούτε θα πρέπει να είμαστε ε, ε, προκατηλημένοι. Άκουσα κάποιες παρεμβάσεις εδώ. υπήρχε αυτή η διάθεση η επεκτατική του συντάγματος που θα ήθελε να συμπεριλάβει και τους Ιούγκρους που δεν διαμένουν στην επικράτεια της Ουγγαρίας. Εμένα μου ήρθε στο μυαλό ο θεμελιώδης νόμος της Βόνης, ο οποίος έλεγε ότι η Γερμανία δεν θα είχε σύνταγμα μέχρι να ενοποιηθεί και να είναι ενωμένοι όλοι οι Γερμανοί. Ήταν ένας επιθυμητός πολιτικός στόχος και επετέχθη αυτό που ήθελαν. Δεν σημαίνει αυτό ότι είχαν υπηρεαλιστικές ε, διαθέσεις οι Γερμανοί τότε. Και θα πρέπει να το δούμε όπως ήταν εκείνη τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Το κυβερνών κόμμα κατά τη διάρκεια της ε, προεκλογικής αναμέτρησης είχε εξηγήσει ότι είχε στόχο να αλλάξει το Σύνταγμα και νομίζω ότι η διέξοδος από τη δικτατορία είναι κάτι που βιώσαμε και στη χώρα μας και η αλλαγή του Συντάγματος εξαιτία της ε, ε, κατάρρευσης της δικτατορίας. Μου άρεσε αυτό που είπε ο κύριος Σάγερ για την ε, συνέχεια που δόθηκε στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει συμπεριληφθεί στο Ουγγρικό Σύνταγμα και σίγουρα αυτό είναι στο DNA των Ευρωπαίων και θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στο Σύνταγμα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Σάγερ διότι ήταν διατεθειμένος να έρθει εδώ να μιλήσουμε και όταν θα έχουμε το κείμενο ενώπιόν μας θα μπορέσουμε να δούμε και τα πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του. Μου άρεσε επίσης και αυτό που ακούσαμε για την δημιουργία μιας επιτροπής η οποία θα μπορούσε να ελέγξει τον προϋπολογισμό εάν ο προϋπολογισμός οδηγούσε σε μεγαλύτερο έλλειμμα. Αυτό είναι καινοτομία. Υπάρχουν και άλλα ε, συντάγματα τα οποία το έχουν συμπεριλάβει στο σύνταγμά τους κατά αντίστοιχο. Ίσως καλό θα ήταν να το μελετήσουμε από πλευράς ε, συνταγματικού δικαίου. Ε, βλέπω κύριε Πρόεδρε ότι θέλετε να με διακόψετε γιατί θέλετε να μιλήσουν και οι υπόλοιποι και θα διακόψω γιατί θυμάμαι ότι θέλετε το λόγο και ο κύριος Μπρόκ. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ στην αρχή σας είπα ότι ήθελα να τελειώσουμε αυτή τη συζήτηση στις 10 γιατί έχουμε πολύ σημαντικές ψηφοφορίες και ότι θα έδινα τις, ε, το λόγο στους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων και στα άλλα μέλη της Επιτροπής μόνο αν υπήρχε άλλος χρόνος. Ακόμα δεν έχει απαντήσει ο κύριος Σέπφλιν, λέει ο πρόεδρος. Έχει ζητήσει το λόγο και ο κύριος Μπρόνς, ο οποίος είναι συντονιστής της ομάδας του. Ε, κατάλαβα, ε, θέλει και το λόγο και ο κύριο Γκουαλτιέρη, αλλά άμα το δώσω σε εσά, πρέπει να το δώσω σε όλου. Αν μου πείτε, ε, υποσχεθείτε ότι θα πείτε μία πρόταση μόνο, συμφωνώ, διαφωνώ, θα σα το δώσω. Αλλιώ, μην ανησυχείτε, θα ξανακάνουμε συζήτηση επί του θέματο. Και η κύρια Γκουρμάη, που είναι αντιπρόεδρος και είναι και αυτή από την Ουγγαρία, ίσως θα έπρεπε να λάβει το λόγο και να μας πει δύο πράγματα. Και εγώ είμαι πρόεδρος, θα μου επιτρέπετε να, να, να πω τίποτα. Αλλά κυρίως θα πρέπει να ακούσουμε και απαντήσεις στις ερωτήσεις που έδεσαν στον κύριο Σάγερ. Ο κύριος Μπρόνς. Μπρόνς. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, είπατε Μπρόνς ή Μπρόκ. Μπρόν, εγώ, πολύ ωραία. Ίσως φαίνεται περίεργη η ερώτηση αυτή, για τους συναδέλφους αυτούς που ε, προέρχονται από χώρες που έχουν ε, συντάγματα. Εγώ μιλάω ερχόμενος από το Νομένο Βασίλειο. Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν όλες αυτές οι αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνθήκη της Λισαβόνας και ιδίως στο ζήτημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην, ε, στο Σύνταγμα αυτό καθ' αυτό. Φαντάζομαι ότι το Σύνταγμα είναι ένα κείμενο πιο αυστηρό και είναι πιο δύσκολο να τροποποιηθεί από την κοινοτική νομοθεσία. Επομένω, θα είναι δύσκολο, πιστεύω πάρα πολύ δύσκολο για την Ουγγαρία να αποσυρθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον, να αποφάσει να κάνει κάτι τέτοιο, ή θα ήταν πολύ δύσκολο ακόμα και να επιβραδύνει τη διαδικασία τη ολοκλήρωση. Ο κύριο ε, Γκουερέρο είπε ότι ε, συνήθως τα συντάγματα υποβάλλονται σε δημοψηφίσματα και ότι ε, δεν θα έπρεπε ενδεχομένω να γίνεται κάτι τέτοιο. Το ξέχασαν όμως αυτό ορισμένα κράτη-μέλη, ιδίως όσον αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας και την έγκρισή της. Γίνανε επίσης κάποιες αναφορές στην Ουγγρική Διασπορά. Δεν έχω εγώ καμία απολύτως αντίρρηση να αναφέρεται το Ουγγρικό Σύνταγμα στην Ουγγρική Διασπορά, γιατί δεν πρόκειται για ανθρώπους που εθελούσια φύγαν από τη χώρα και εγκατέλειψαν τη χώρα τους και πήγαν να ζήσουν σε μια άλλη χώρα. Είναι άνθρωποι που είναι θύματα της ε, ε, συνθήκης του 1920 που αφαίρεσε από την Ουγγαρία ένα πολύ μεγάλο τμήμα από την επικράτειά της. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη από τους υπολείπους, ε, στους οποίους δεν θα δώσω τους λόγους γιατί έχει πάει σχεδόν 10 και 10 θα ήθελα να δώσω στην κυρία Γκουρμάη το λόγο, αλλά σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ακούσαμε ότι το Σύνταγμα αυτό κρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία και σωστό είναι και χτες το κόμμα Φίντες έδωσε τις ευλογίες σε αυτό το σχεδόν μονοκομματικό Σύνταγμα. Τώρα όμως θα πρέπει να υπάρξουν και νομικές εγγύησεις. Ισχυρίστηκε ο μιλητής ότι έγινε μεγάλη διαβούλευση και οι πολίτες υποστήριξαν, λέει, το Σύνταγμα. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Κάτι πάει στραβά και εδώ, γιατί από το παλιό Σύνταγμα έχουμε ένα κανόνα που λέει ότι για να ψηφιστεί ένα νέο και να γίνει αναθεώρηση ή να έρθει ένα νέο σύνταγμα χρειάζεται πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων της Βουλής. Και μας είπαν ότι εντάξει μπορούσε να έχει κάνει τροπολογίες και η αντιπολίτευση. Βέβαια, δεν την άκουσαν την αντιπολίτευση, ούτε στις συνεδριάσεις που έγιναν ούτε όταν έλεγε τη γνώμη της. Ούτε καν τον πρόεδρο του συνταγματικού δικαστηρίου δεν άκουσαν. Μας είπαν ότι έστειλαν ένα εκατομμύριο απαντήσεις οι πολίτες. Ήταν 12 ερωτήσεις, αλλά το διάστημα που είχαν τη ε, στη διάθεσή τους να απαντήσουν οι Ούγγροι πολίτες ήταν 15 μέρες, ίσως και λιγότερο αυτό δεν είναι δημοσκόπηση, δεν είναι δημοψήφισμα ούτε διαβούλευση με τον πληθυσμό. Και λιγότερο από ένα τρίτο του πληθυσμού απεφάνθη για το Σύνταγμα. Ουσιαστικά για τα μάτια ήταν και το ερωτηματολόγιο, προφάσεις. Αντί να γίνει πραγματική εθνική δημόσια διαβούλευση, έστειλαν ένα ερωτηματολόγιο. Και για να έρθει νέο σύνταγμα χρειάζεται δημοψήφισμα. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ακούσαμε και χτες μετά την τελική ψηφοφορία. Το έγραψαν και οι διεθνείς εφημερίδες, ο Φιγκαρό, οι Financial Times και οι γερμανικές εφημερίδες που έλεγαν ότι είναι το πρώτο σύνταγμα μιας αυταρχικής κυβέρνησης στην Ευρώπη, το πρώτο αυταρχικό σύνταγμα της Ευρώπης. Χάθηκαν τα δικαιώματα των συνδικάτων, τα δικαιώματα τα κοινωνικά, των εργαζομένων, τώρα δεν μπορώ να πω και στις λεπτομέρειες. Κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι το Σύνταγμα είναι πραγματικά ο θεμελιώδης νόμος για ένα κράτος, για τη λειτουργία του. Εχθές λοιπόν εγκρίθηκε αυτό το Σύνταγμα, αλλά ε, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι αυτό μόνο η αρχή μιας νέας συντακτικής διαδικασίας, για να έχουμε εκτός από Σύνταγμα και δημοκρατική νομιμότητα. Αυτό θα το αλλάξουμε. Λοιπόν, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε στο πλευρό μας και το λαό και την κοινωνία συνενετικά ένα ειλικρινές και τίμιο σύναγμα για τη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη εκ νέου από τους συναδέλφους που δεν μπορώ να τους δώσω το λόγο. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Σάγερ, επειδή αναφέρθηκαν όλοι στην εθνική τους εμπειρία, θα ήθελα να πω και δύο πράγματα για την ιταλική εμπειρία που έχει ένα πολύ σταθερό σύνταγμα από το 1948 και η παρούσα κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα ήθελε να αλλάξει ε, αλλά δεν νομίζω και δεν ελπίζω ότι θα αλλάξει. Και να σας πω ότι το Σύνταγμα αυτό ψηφίστηκε μετά από ένα δημοψήφισμα για την ε, πάυση της μοναρχίας, αλλά είχαμε και συντακτική συνέλευση και μια νομοθετική διαδικασία για το Σύνταγμα. Και θα ήθελα να ξέρω εάν στη διάρκεια της, προεκλογική της προεκλογικής εκστρατείας παρουσιάστηκε στο εκλογικό πρόγραμμα του κόμματος που κέρδισε τις εκλογές ένα σχέδιο τροποποίησης του Συντάγματος ώστε να μπορούμε να μιλάμε και για μια συντακτική συνέλευση ουσιαστικά. Ε, ευχαριστώ τον κύριο Σάγκερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ε, μου δίνετε τη δυνατότητα να συμμετέχω στην ε, διαδικασία αυτή. Στην αρχική μου παρέμβαση δεν μπόρεσα να μιλήσω πάρα πολύ για τη διαδικασία, αλλά στο ζήτημα αυτό αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι. Επομένω, θα ήθελα να πω ότι η Ουγγαρία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νέο σύνταγμα τα τελευταία 20 χρόνια. Ε, το σύνταγμα το οποίο υφίσταται ακόμα αυτή τη στιγμή είναι το, το, το προηγούμενο μας σύνταγμα. Το σημαντικό ήταν να καταφέρουμε να πετύχουμε μία συνένεση. Δεν είχαμε καταφέρει από όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν από τον κομμουνισμό μέχρι σήμερα να καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα νέο σύνταγμα και το πετύχαμε αυτό χθε. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι δεν ήταν μόνο τα μέλη του Κοινοβουλίου αλλά το γενικότερο κοινό το οποίο συμμετείχε στην όλη διαδικασία διαμόρφωσης του συντάγματος. Η κυρία Τζίτα Γκουρμάη έκανε μία δήλωση, δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αναφερθώ σε αυτήν, να απαντήσω σε αυτήν, δεν θα ήθελα να φέρω την εσωτερική συζήτηση που γίνεται στη χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το δικό τη όμω το κόμμα είχε τη δυνατότητα να πει ό,τι ήθελε να πει στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο, αλλά αποφάσισαν να μην το κάνουν. Αυτό αποφάσισαν να μην εκπροσωπηθούν, να μην εκπροσωπήσουν του ψηφοφόρου του στην συνταγματική διαδικασία, στη διαδικασία σύνταξη του συντάγματο. Δική του επιλογή ήταν αυτή. Δεν θα ήθελα πάντω να φέρθω περισσότερο σε αυτό. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, επομένω θα ήθελα να πω στου συναδέλφου ε, ότι μπορώ να απαντήσω σε επιμέρου σημεία τα οποία έθιξαν, ωστόσο θα ήθελα να κάνω κάποιε γενικέ παρατηρήσει. Πρώτον, εκτιμώ ιδιαίτερα το γνήσιο ενδιαφέρον το οποίο δείχνεται για το Σύνταγμά μα. Θεωρώ ότι έτσι θα πρέπει να διεξάγονται τα πράγματα ανάμεσα σε διαφορετικά έθνη και κράτη τα οποία ε, ενωμένα κινούνται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές ε, συνταγματικές παραδόσεις. Επομένως είναι περίεργο για μένα να ακούω ότι ένας Γερμανός ε, πολίτης ζητά να διεξαχθεί ένα δημοψήφασμα σε μια χώρα που δεν προβλέπει κάτι τέτοιο σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι από το Βέλιο, για παράδειγμα που την προηγούμενη εβδομάδα είπαν το σταγματικό δικαστήριο στην... για το συνταγματικό δικαστήριο στην Ουγγαρία και έγινε το σχόλιο αυτό από μια χώρα που δεν έχει συνταγματικό δικαστήριο. Έχετε ενδεχομένω εσεί κάποιο άλλο διαφορετικό σύστημα εκτό μικροφώνου η παρέμβαση του κ. Φερχόφστατ. το μόνο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε διαφορετικές συνταγματικές παραδόσεις. Η Ουγγαρία τα τελευταία χίλια χρόνια κατάφερε να δημιουργήσει μια πολύ καλή συνταγματική παράδοση η οποία παρουσιάζει τις δικές μας τις ιδιαιτερότητες. Στο πλαίσιο λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μαθαίνουμε ημένα από του ΔΕ, παρακολουθούμε πολλέ φορέ τα παραδείγματα των άλλων κρατών. Αυτό που θα ήθελα πάντω να αποσαφηνίσω είναι ότι το κείμενο, το τμήμα αυτού του κειμένου είναι διαθέσιμο, έχει εδώ και κάποιε εβδομάδε, δεν έχει τροποποιηθεί πολύ και αναφερόμαστε στο σύνολο των ε, δικαιωμάτων. Δεν υπάρχουν ε, δικαιώματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο στο κείμενο. Θα ήθελα λοιπόν να διαβάσετε το κείμενο, αυτό το οποίο δεν έχει τροποποιηθεί. Πρόκειται ουσιαστικά για την ε, κοινή κληρονομιά που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα δικαιώματα. Δεν έχει τροποποιηθεί λοιπόν το κείμενο αυτό. Υπάρχουν όμω από την άλλη, όπω είπαμε, διαφορετικέ παραδόσει ω προ το Σύνταγμα. Ορισμένοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο ζήτημα του δημοψηφίσματο. 23 νέα συντάγματα εγκρίθηκαν τελευταία 20 χρόνια στην Ευρώπη μόνο για δέκα από αυτά έγινε δημοψήφισμα. Επίσης αναφερθήκατε στους δικαστές. Υπάρχουν πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ανάλογες διατάξεις όπως και το δικό μας το Σύνταγμα όσον αφορά το όριο ηλικία για τις συνταξιοδότηση και σε καμία περίπτωση αυτό δεν εισάγει κάποια διακριτική μεταχείριση. Δεν μπορώ να καταλάβω το επιχείρημα αυτό. Ισχύει όπως σας είπα αυτό το όριο ηλικία και σε πολλές άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαθαίνουμε λοιπόν μένουν από τους ΔΕ, μαθαίνουμε από την εμπειρία άλλων κρατών και έχουμε παράλληλα και τη δική μας την παράδοση. Για παράδειγμα, πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στους Ούγγρους που ζουν στο εξωτερικό. Μα δεν πρόκειται για κάποια αλλαγή που γίνεται στο Σύνταγμα. Υφίσταται και στο νυν Σύνταγμα. Λέμε ότι η Ουγγαρία αναλαμβάνει ευθύνη για τους Ούγγρους που ζουν στο εξωτερικό προκειμένου να καταφέρουν αυτοί να διατηρήσουν την κοινωνική του ζωή, την εθνική τους παράδοση και τον εθνικό τους πολιτισμό. Πρόκειται για μια υποχρέωση του κράτους προς τους ανθρώπους αυτούς και σε καμία περίπτωση δεν έχει κάποια αλυτρωτική διάσταση. Επίσης, όσον αφορά τη θανατική ποινή, ξέρετε ότι έχουμε ένα σταγματικό δικαστήριο το οποίο έχει απαγορέψει τη θανατική ποινή. Αυτό αποτελεί τμήμα του δικαστικού μας συστήματος. Και όπως ξέρετε έχουμε προσυπογράψει διεθνείς συνθήκες ως προς αυτό. Και αυτό ισχύει επίσης και για τη διακριτική μεταχείριση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε ότι ε, ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν είναι κάτι το οποίο απουσιάζει από το νομικό σύστημα της Ουγγαρίας. Η Ουγγαρία έχει προσχωρήσει σε διεθνείς συνθήκες, αποτελεί αυτό το τμήμα της νομοθεσίας μας και έχουμε ουσιαστικά διατηρήσει το κείμενο το οποίο υπάρχει τα τελευταία 20 χρόνια και που έχει να κάνει με τις διακρίσεις αυτές, με την καταπολέμηση των διακρίσεων. Άλλωστε, οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων απαγορεύεται από το σύνδειγμά μας. Ακόμα και στο τέλος του κειμένου λέγεται και άλλες μορφές διάκρισης. Επομένως όσοι έχουν ανησυχίες ως προς αυτό δεν έχουν παρά να δούνε πώς λειτουργούν τα πράγματα στην πράξη. Είμαστε μια δημοκρατική χώρα με δημοκρατικούς θεσμούς, με σταγματικό δικαστήριο. Τα δικαιώματα αυτά υφίστανται, προασπίζονται και μπορεί να γίνουν προσφυγές στα δικαστήριά μας κάθε φορά που υπάρχει μια καταπάτηση. Οποιαδήποτε διάκριση απαγορεύεται σύμφωνα με το νυν ουγγρικό ε, νόμο, δίκαιο και αυτό άλλωστε λέει, άλλωστε, αυτό λέει και το νέο κείμενο του συντάγματος. Όσον αφορά τα δικαιώματα του Προέδρου, μα ο Πρόεδρος πάντα είχε το δικαίωμα αυτό. Δεν λέμε ότι θα καθορίζουμε εμεί ευρωπαϊκές εκλογές σε διαφορετική χρονική περίοδο από τις άλλες χώρες. Πάντως και το νυν σύνταγμα αναφερόταν σε αυτό το δικαίωμα του Προέδρου όσον αφορά τον καθορισμό της χρονικής περίοδου των εκλογών. Όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα σας διαβεβαιώ ότι ε, υπάρχει σαφώς, αναφέρεται σαφώς το δικαίωμα της απεργίας. Είναι από τα λίγα εθνικά συντάγματα που αναφέρεται στην πλήρη απασχόληση δεν λέει ότι ε, ο πολίτης έχει το δικαίωμα να εργάζεται σε μια θέση απασχόλησης που ε, παρέχει το κράτος. Λέει ότι το κράτος θα πρέπει να δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες όποιος επιθυμεί να δουλέψει θα μπορεί να το πράξει, θα μπορεί να εργαστεί. Επομένως όλες αυτές οι ανησυχίες για το αν αντικατοπτρίζονται σωστά τα δικαιώματα, οι αξίες, οι αρχές, οι ανησυχίες αυτές λοιπόν δεν είναι βάσιμες και θα σας, μάλλον σας αποστήλαμε και το κείμενο πριν από τρεις-τέσσερις εβδομάδες. Σας καλώ να το διαβάσετε. Ξέρετε ότι πολλοί είμαστε νομικοί, νομομαθείς, κάθε λέξη έχει την έννοιά της και για πρώτη φορά ουσιαστικά αναφερόμαστε εδώ πέρα στα συνταγματικά δικαιώματα πολύ περισσότερο από ό,τι σε προηγούμενα κείμενα του Ουγγρικού Συντάγματος. Εμένουμε λοιπόν στα σημεία αυτά και θεωρούμε ότι το νέο Σύνταγμα αποτελεί μια βελτίωση. Το ζήτημα τώρα της νομιμότητας. Ναι, προφανώς η Ουγγαρία είναι μια δημοκρατία, γίνονται συζητήσεις ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Η νομιμοποίηση όμως σύμφωνα, σύμφωνα με το Ουγγρικό Σύνταγμα προβλέπεται μέσω των εκλογών. Υπάρχουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών που λειτουργούν στα πλαίσια της κυβέρνησης και εξουσιοδοτούνται να διαπραγματεύονται το Σύνταγμα. Και δημιουργήθηκε μία επιτροπή ήδη από τον Ιούνιο πέρυσι, όπου προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν όλα τα πολιτικά κόμματα για τη διαμόρφωση του τελικού συνταγματικού κειμένου. Η όλη διαδικασία λοιπόν ήταν ιδιαίτερα διαφανής και ουσιαστικά υπερβαίνει τα όρια του Εθνικού μας Κοινοβουλίου και είχαμε προβλέψει και νέους τρόπους συμμετοχής των πολιτών. Είχαν, γίνανε έρευνε, ένα ερωτηματολόγιο με 12 ερωτήσει, ενδεχομένω να πείτε ότι αυτό δεν αρκούσε. Μόνο και μόνο το να συμπληρώσει κανείς το έντυπο αυτό με τις 12 ερωτήσεις απαιτούσε περίπου μισή ώρα από τους πολίτες. Η κυρία Γκουρμάη είπε ότι ε, δεν ε, διεξήχθη σωστά τη διαδικασία αυτή. Εγώ όμω ε, παρακολούθησα πραγματικά τη διαδικασία αυτή. Μπόρεσε να συμμετάσχουν, μπόρεσε να συμμετάσχουν όντως οι πολίτες και τα πράγματα κινήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε όσο, όσο δυνατόν περισσότερους πολίτες γινότανε. Ξέρετε ότι το 1989 όταν έγινε η μετάβαση προς τη δημοκρατία δεν υπήρχαν τότε εκλεγμένα κόμματα δεν υπήρχε σωστή εκπροσώπηση. Η εκπροσώπηση δεν ήταν απόλυτα νομιμοποιημένη. Επομένως ήταν πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα νέο σύνταγμα το οποίο θα εκπροσωπεί περισσότερο τους πολίτες, αναφέρεται στις βασικές αρχές της δημοκρατίας και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά κύριε Πρόεδρε, που μου δώσετε τη δυνατότητα να ενημερώσω για το νέο μα αυτό σύνταγμα του συναδέλφου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφύγουμε οποιαδήποτε παρανόηση και αυτό θα το πετύχουμε μόνο αν δίνουμε αυτή την κατάλληλη ενημέρωση και αν διασκεδάζουμε οποιαδήποτε αμφιβολία και ανησυχία μπορεί να υπάρχει. Ακόμα και μετά το τέλο τη τη αυτή, είμαι στη διάθεσή σα για να σα δώσω περαιτέρω πληροφορίε. Φαντάζομαι ότι ξέρετε το κείμενο ήδη πολύ καλά. Θα μπορούσα να σα δώσω όμω κάποιε περαιτέρω εξηγήσει, αν τυχόν έχετε ανησυχίε ή αμφιβολίε για το κείμενο αυτό. Είμαι στη διάθεσή Είμαι ο συναδελφό σα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι σε θέση να σα δώσω αυτέ τι πληροφορίε. Είναι σημαντικό να έχουμε και εμεί μια δημοκρατική συζήτηση για τα συντάγματά μα. Και ουσιαστικά μια τέτοια συζήτηση προποθέτει ότι θα πρέπει καταρχά να καταβάλουμε περί τίνο πρόκειται το όλο εγχείρημα και στη συνέχεια να μιλήσουμε για πολιτικέ συζητήσει ή για πολιτική αντιπαράθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οποιαδήποτε ζήτηση κάνουμε να βασίζεται σε σωστές και κέρυες πληροφορίες. Και είμαι σίγουρος ότι τις πληροφορίες αυτές θα είμαι σε θέση να τις δώσω εφόσον το επιθυμούν οι συναδελφοί μου στα πλαίσια της εξαιρετικής αυτής επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζάγερ. Αναμένουμε και το κείμενο μεταφρασμένο. Εν τω μεταξύ έχουμε σημειώσει όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε, οι οποίες ναι μεν ήταν συνοπτικές αλλά πλήρεις. Να περάσουμε ε, πολύ γρήγορα στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης. Έχουμε να ψηφίσουμε δύο εκθέσεις. Η πρώτη έκθεση είναι του συναδέλφου Ντάφ ε, για την τροποποίηση της πράξης του 1976. Σας έχω ζητήσει να φέρετε και τις ε, κάρτες σας, γιατί μπορεί να χρειαστεί σε πολλές περιπτώσεις νομίζω να κάνουμε και ηλεκτρονική επαλήθευση. Ε, λοιπόν, την, ε, τις κάρτες σας μπορούμε να ξεκινήσουμε να ψηφίσουμε. Κύριε Ντάφ, ψηφίζουμε αμέσω. Ωραία, τέλεια. Να ξεκινήσουμε με ανάταση χειρός και μετά βλέπουμε. Άρθρο 14, παράγραφος 2, συμβαστική τροπολογία α του εισηγητή. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται και με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Θεωρούμε λοιπόν ότι καλύπτονται από το συμβιβασμό όλες οι ε, τροπολογίες που έχουμε στη συνέχεια. Έχετε τις τροπολογίες άλλωστε ενώπιον σας. Μπορώ να σας πω σε ποια σελίδα πηγαίνουμε. Μέχρι τη σελίδα 4 λοιπόν. Τροπολογία Β του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και πάλι στο άρθρο 7, τροπολογία 104 καταπίπτει γιατί ψηφίστηκε η τροπολογία, υπερψηφίστηκε η τροπολογία Β, όπως επίσης και η 105 και η 106. Περνάμε τώρα στο άρθρο 8, τροπολογία C του εισηγητή, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει η 107. Τροπολογία D του εισηγητή. Δεν καταπίπτει. Όχι. Ψηφίζουμε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 108 καταπίπτει. καταπίπτει γιατί ψηφίσαμε την D, το ίδιο ισχύει και για την 109 και την 110. Τροπολογία 1 του εισηγητή, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 2, 111, Σμιτ, υπέρ, παρακαλώ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στο άρθρο 2α νέο, συμβιβαστική τροπολογία β του εισηγητή. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 2, 112, 115, 117, 118, 116, 113, 114 και περνάμε στη συμβαστική τροπολογία L στη σελίδα υπαριθμών 8. Α, το λόγο. Κύριε Γουαλτιέρη, θέλετε το λόγο. Ναι, ήθελα να προτείνω μία προφορική τροπολογία στη συμβαστική τροπολογία L να αντικαταστήσουμε την αναφορά μέθοδο Sant League στη μέθοδο Don't. Ο εισηγητής. Ε, ε, Κύριε Πρόεδρε, δεν συμφωνώ με την προφορική εφητροπολογία. Δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Είναι κάποιος αντίθετος. Κύριε Πρόεδρε, είναι βασική αυτή η πληροφορία. Θα μπορούσε να γίνει ηλεκτρονικός ε, η επαλήθευση της τροπολογίας. Ah, λοιπόν, ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία L. Ζητήθηκε ηλεκτρονική επαλήθευση.

Non, sinistra. A sinistra, credo. No, no, scusate, questo, il voto è come in aula, quindi il sì a sinistra e... Lipon. Λοιπόν, είναι ναι αριστερά, όχι δεξιά και στη μέση αποχή. Εύκολο μπορείτε να ψηφίσετε. Ψήφισαν όλοι, ωραία, πέρασε ψηφοφορίας. ψηφοφορία. 19 υπέρ, 3 κατά, 22 ψηφίσαντες, καμία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν. Επομένως, πηγαίνουμε απευθείας στην τροπολογία 4 του εισηγητή και 121 Βίλαν στην παράγραφο 1 που είναι πανομοιότυπες υπέρ Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν για τις τροπολογίες 4 του εισηγητή και 121 βίλαν που είναι πανομοιότυπες. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 9 υπέρ, 10 κατά μία αποχή απορρίπτεται. Προχωράμε λοιπόν. Τροπολογία Γκουαλτιέρη 122. 122 έχω εγώ εδώ. Δεν καταπίπτει γιατί δεν εγκρίθηκαν οι 421. 122 υπέρ για την ε, τροπολογία Γκουαλτιέρη. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2 νέα έχουμε τις τροπολογίες 4 και 122 πανομοιότυπες υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίζουμε την τροπολογία και 122 που είναι πανομοιότυπες. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 14 υπέρ, 8 κατά, εγκρίνεται. Περνάμε στην 121 Βίλαντ, η οποία όμως ε, καταπίπτει διότι εγκρίθηκαν οι 422, 123 γκουαλτιέρι. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5 του εισηγητή, πανομοιότυπη με 124 Βίλαντ. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Και πάλι την ίδια πλειοψηφία με πριν εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην 124. Ράινερ Βίλαντ η οποία καταπίπτει. Τροπολογία 6 του εισηγητή στο άρθρο 5. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 125 Γουαλτιέρη. Υπέρ Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 126 Βίλαντ. Υπέρ. Κατά. Και πάλι η ίδια εγκρίνεται. Τροπολογία 8 καταπίπτει. 127 καταπίπτει επίσης. 128 επίσης. 129 Πρέπει να ψηφίσουμε την 128 γιατί απορρίφθηκε 125. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 129. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 και πάλι το εισηγητή. Υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία C στο άρθρο 9 της εισηγητή υπέρ κατά αποχές δίνεται που σημαίνει ότι καταπίπτουν καλύπτονται μάλλον από την τροπολογία οι 11 και οι 130 και φτάνουμε Στη συμβαστική τροπολογία D, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία D, που καλύπτει τις 131 και 12 του εισηγητή. Είμαστε τώρα στην τροπολογία 13 του εισηγητή. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 που καταπίπτει μερικός εάν απορριφθούν ε, κάποιες τροπολογίες αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο επομένως ψηφίζουμε τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 16 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 132 καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε 16. 17 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 η οποία καταπίπτει γιατί εγκρίθηκαν ο συμβασμός Α και L. 133 Η 18 Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Ντάφ, ζητώ συγγνώμη. Πρέπει να ψηφίσουμε τη 18. Λέει, καταπίπτει εάν οι συμβιβασμοί απορριφθούν. Αλλά οι συμβιβασμοί υπερψηφίστηκαν. Επομένως, πρέπει να ψηφίσουμε τη 18. Α, ναι, έχετε δίκιο. <laughs> Συγγνώμη. Ψηφίζουμε λοιπόν το 18 της εισηγητή. Υπέρ. elettronico? 11, 12. Να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 13 υπέρ, 10 κατά. Εγκρίνεται. Κατόπιν. Τροπολογία 133, η οποία όμως καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε η 18. Τροπολογία 19 του εισηγητή, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καλύπτονται λοιπόν οι 134 και οι 20 των Γουαλτιέρη και του εισηγητή, τροπολογία 21 του εισηγητή. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 22 και πάλι του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 23, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 135 η οποία καλύπτεται από τον συμβιβασμό Β, το ίδιο και η 136 και η 137 και η 138. Πρέπει τώρα να ψηφίσουμε την 62 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 63. Υπέρ. Κατά. Και πάλι η διαπλειοψηφία Απορρίπτεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65. Η 66. Η 67 και η 68 καταπίπτουν. 69 επίσης η 70 πρέπει να την ψηφίσουμε Ψηφίσουμε λοιπόν την τροπολογία 70 υπέρ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 Ah, ah, η κυρία Γκουρμάη θέλει να κάνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Ωραία λοιπόν. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 70. Άρχεται η ψηφοφορία. η ψηφοφορία. 16 υπέρ, 6 κατά. 71. Καταπίπτει. 72. Επίσης. 73. Τροπολογία Σόλτς. Ψηφίζουμε υπέρ. Abbiamo votato il 73. Ηλεκτρονική e, e επαλήθευση για την 73. παράγραφο 2 Σόλτς. Η... Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. 13 ψήφοι υπέρ, 10 κατά. Εγκρίνεται. 74. κατά καταπίπτει. Συμβιβαστική τροπολογία F του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 75, η οποία καλύπτεται από τη συμβιβαστική τροπολογία F. Δεν ψηφίζουμε λοιπόν. Όπως επίσης και η 76, 77, 78, 79 και φτάνουμε στην 80. Άλιν Σμιτ για την παράγραφο 3α. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 81 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82 Χάγκλουντ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία G του εισηγητή. Sì, sì, 82 abbiamo Συμβαστική τροπολογία G για την παράγραφο 4. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την συμβαστική τροπολογία G. Άρχεται η ψηφοφορία. Chiudo la votazione. Πέραση ψηφοφορία. 16 υπέρ, 7 κατά εγκρίνεται. Επομένως, μπορούμε να περάσουμε τις 83 και 84 που καλύπτονται και πάμε στην 85 και 86 τις οποίες θα ψηφίσουμε από κοινού για την παράγραφο 5. Υπέρ παρακαλώ. Και κοντράριο. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 86. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 10 voti 13 ψήφοι 13 κατά. Συμβαστική τροπολογία age του εισηγητή. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 16 ψήφοι κατά, 5 υπέρ, μία αποχή. Τρίτο τμήμα, όρος ethnic. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τρίτο και τελευταίο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 88 καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία όπως και 87. 89. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 90. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 91. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. 91 Χέφνερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 14 ψήφοι υπέρ, 9 κατά. Παράγραφος 6. Τροπολογία, ε, προφορική τροπολογία. Τροπολογία 92 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93 Βίλαντ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 94 αποσύρεται 95 και 96 μαζί υπέρ κατά απορρίπτεται 97 Καταπίπτει γιατί εγκρίθηκαν οι τροπολογίες 1-24. Συμβαστική τροπολογία ΑΗ του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καλύπτεται 27. Ψηφίζουμε την 28. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 29 Γκουαλτιέρη υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 30 και πάλι γουλτιερή πέρ κατά νομίζω ότι απορρίπτεται να κάνουμε όμως μια επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 30 γκουαλτιέρη άρχεται η ψηφοφορία πέρες ψηφοφορίας Απορρίπτεται 15 ψήφοι κατά 9 υπέρ. 31 γκολτιέρ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται νομίζω. 32. Θέλετε να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. 31 λοιπόν. 31 ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. È chiusa la votazione. 12, 12. Eh, non è approvato perché siamo 12. 12 per 12 κατά απορρίπτεται. Καλώ επαληθεύσαμε. Τροπολογία 32 γκολτιέρι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Επαλήθευση και πάλι. 32 Γουαλτιέρη. Άρχεται η ψηφοφορία. η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 14 ψήφοι υπέρ, 9 κατά, μία αποχή. Καταπίπτει 33, γιατί εγκρίναμε τη 32, 34 σέπφλιν υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 35 γκουαλτιέρι υπέρ κατά απορρίπτεται. 36 αποσύρεται. 37 γκουαλτιέρι υπέρ κατά απορρίπτεται. 38 Οι 38 και 39 είναι πανομοιότυπες. Δεν θα τις ψηφίσουμε. Δεν είναι ουσιαστικό το πρόβλημα, είναι θέμα μετάφρασης, δεν τις ψηφίζουμε. 40. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41 καταπίπτει, γιατί εγκρίθηκε η 40. 42 υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. 43 κατά όχι. Ψηφίζουμε. Υπέρ για τη 43 παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω, αλλά να κάνουμε και μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 12 υπέρ, 11 κατά. Μία εποχή. Τροπολογία 44 Γουαλτιέρη υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. 44 γκολτιέρι. Άρχεται η ψηφοφορία. Εκείουσα votazione. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 16 ψήφοι κατά 6 υπέρ. Συμβαστική τροπολογία J. Ακριβώς το Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, Ηλεκτρονική επαλήθευση, δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ε, Απορρίπτεται. 8 ψήφοι υπέρ, 16 κατά. Καλύπτονται οι 45, 46, 47, 48, 49. Πηγαίνουμε στην 50. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 51 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 52 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 53, 54 και 55 είναι πανομοιότητες, τις ψηφίζουμε από κοινού, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται 56 υπέρ κατά απορρίπτεται 57 υπέρ κατά εγκρίνεται η 58 μισό λεπτό να ελέγξουμε καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία Α και από άλλες, επομένως δεν ψηφίζουμε. Συμβαστική τροπολογία K του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 59 καλύπτεται και η 60 καλύπτονται από άλλο συμβιβασμό. Τροπολογία 61, Γουαλτιαρή υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Επαλήθευση. Ωραία. Τροπολογία 61. Αιτιολογική σκέψη Z. Άρχεται η ψηφοφορία. θα να βοηθάξω. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 15 ψήφοι υπέρ, 7 κατά. Δύο αποχές. Τροπολογία 25 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τελική ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως τροποποιήθηκαν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη Εγκρίνεται. 20 ψήφοι υπέρ, 4 κατά. Συγχαρητήρια κύριε Νταφ, ε, ειλικρινώ αυτή τη φορά. Ο οποίο έδωσε αίσιο τέλος σε μια επιχείρηση η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για τις δύο επόμενες εκθέσεις. Η μία έχει να κάνει με τη διοργανική συμφωνία σχετικά με ένα κοινό μητρό διαφάνειας. Ξεκινάμε λοιπόν με την έκθεση αυτή.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 Ξεκινάμε με την έκθεση για τη διοργανική συμφωνία σχετικά με ένα κοινό μητρό διαφάνειας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Εγώ είμαι ο συγητής. Ψηφίζουμε λοιπόν. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Ο κύριος Χέφνερ. Ναι, συγγνώμη που ζητώ το λόγο. Μετά τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, επιθυμώ να αποσύρω την παρούσα τροπολογία, δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. Η 32 λοιπόν αποσύρεται. Περνάμε στην τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται 34. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση όμως για την 34 θα κάνουμε τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 16 υπέρ, 7 κατά. Τροπολογία παριθμών 3 Μέλτσερ υπέρ. Κατά. ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 3 Μέλτσερ, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 14 υπέρ 9 κατά. Τροπολογία DAF. Για την τροπολογία αυτή ζήτησα να γίνει ψηφοφορία σε ξεχωριστά τμήματα το πρώτο τμήμα καταπίπτει, επομένως θα ψηφίσουμε το δεύτερο και το τρίτο τμήμα μόνο. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα το, ελέγξουμε, ηλεκτρονικά. Το τρίτο τμήμα της τροπολογίας υπαριθμών 1 του κυρίου Νταφ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται για μία ψήφο. Τροπολογία 2 Μπέρμαν που καλύπτεται από την τροπολογία υπαριθμών 1. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 4, Μπέρμαν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 6, Μόλτσερ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 5, Πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 5. Θέλετε, κύριε Χέφνερ, να την αποσύρετε. Θέλετε να αποσύρετε την τροπολογία αυτή. Όχι. Την ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 7, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 για τερμάνκι θα μπορούσε να συνδυαστεί με την τροπολογία 9. Τις ψηφίσουμε και τις 2. Υπέρ τις 10. Κατά. Εγκρίνεται. Μπέρμαν υπαριθμών 9. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 8. Γκρόιτε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία α. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε τις 11, 12, 13, 14, 15, εγκρίθηκε η συμβαστική τροπολογία α, επομένως καταπίπτει η τροπολογία 16, περνάμε, καλύπτουμε τις 17 και τις 18 και την 19, καταπίπτει και η τροπολογία 20, γιατί ψηφίστηκε η συμβαστική τροπολογία Β, επομένως πρέπει να ψηφίσουμε τροπολογία 21. Σέντεργαρτ, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται 22. Υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Το πρώτο τμήμα της 24 καλύπτεται από τη συμβαστική α, το δεύτερο τμήμα δεν το ψηφίζουμε δεν είναι παραδεκτό. Δεν ψηφίζουμε την 25, 26, 27 γιατί καλύπτονται από τη συμβαστική Α και Σ. 28 δεν την ψηφίζουμε γιατί το πρώτο τμήμα καλύπτεται από τη συμβαστική Α, το δεύτερο τμήμα δεν είναι παραδεκτό γιατί ζητά την τροποποίηση συμφωνίας 29 Μπέρμαν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 Ντάφα υπέρ κατά, εγκρίνεται. 35 Σάντεργκαρτ υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 37 δεν είναι παραδεκτή γιατί ζητά τροποποίηση της συμφωνίας δεν είναι δυνατό, 38 δεν είναι παραδεκτή γιατί για μία ακόμη φορά ζητά την τροποποίηση της συμφωνίας που δεν είναι δυνατό βέβαια να γίνει κάτι τέτοιο. Τελική λοιπόν ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία, πέρας. Ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα, 22 υπέρ, ουδής κατά. Ας περάσουμε τώρα στην τελευταία έκθεση που πρέπει να ψηφίσουμε, τροποποίηση του καονισμού μετά τη θέσπιση ενός κοινού μητρώου διαφάνειας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Ξεκινάμε με το άρθρο Μητροπολογία 13 Μπέρμαν υπέρ Τροπολογία περιθμών 13 για το άρθρο 9 από τον κύριο Μπέρμαν. Υπάρχει μια κάποια σύγχυση. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία περίθμων 13 Μπέρμαν άρχιτη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 19 υπέρ 3 κατά. Δεν θα ψηφίσουμε την τροπολογία 1. Τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά. Η τροπολογία 3 έχει αποσυρθεί. Περνάμε στην 14 υπέρ. κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 15

No, detto di votare sì, tutto. Mm? Quindi raccomanderei di non votare per... Eh, Δεν θα ψηφίσουμε κατά τμήματα, σας προτείνω να ψηφίσουμε το σύνολο της τροπολογίας αυτής. Εκτός κι αν κάποιος εμένει για ψηφοφορία κατά τμήματα για την τροπολογία 15, όχι λοιπόν, ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά απορρίπτεται. Εγκρίνεται, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. 9 υπέρ κατά εγκρίνεται. 10 δι υπέρ κατά εγκρίνεται. 11D υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 17 δεν είναι παραδεκτή γιατί ζητά τροποποίηση που δεν μπορούν να γίνουν. 12 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 23 υπέρ. Ομόφωνα εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ και ολοκληρώνεται κατά αυτόν τον τρόπο η ψηφοφορία. Να περάσουμε λοιπόν τώρα. Abbiamo... 11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 Λοιπόν, έχουμε ακόμα μία γνωμοδότηση, την έκθεση Σαουντάργα εδώ. Επειδή απουσιάσω για 10 λεπτάκια, θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Τσαρκόσκι να αναλάβει εδώ τα ενία για τη συζήτηση της γνωμοδότησης Σαουντάργας, που είναι το τελευταίο θέμα που έχουμε στη μερίσια διάταξη πριν από την ε, παρουσία εδώ του κυρίου Τρεμόντι. Uh, Ας περάσουμε τώρα στην γνωμοδότηση για την Επιτροπή Προπολογισμών. Το λόγο έχει ο συντάκτης γνωμοδότησης, ο κύριος Σαουντάγκρας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση που δεν διαφέρει πολύ από αυτήν που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ο προπολογισμό δεν πρόκειται να αυξηθεί ιδιαίτερα και δεν νομίζω ότι θα έχουμε και σημαντικές περικοπές όμως από την άλλη. Συνεπώς, η θέση μας φέτος ομοιάζει πάρα πολύ με αυτή που είχαμε πέρυσι. Αναφερόμαστε σε ζητήματα τα οποία εξακολουθούν να μας απασχολούν. Ωστόσο η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να λάβουμε υπόψη νέες αλλαγές, νέες εξελίξεις. Ο κανονισμός για την πρωτοβουλία των πολιτών έχει τεθεί σε ισχύ και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πλήρως από την 1η Απριλίου του 2012. Στη γνωμοδότησή μου λοιπόν αυτή τονίζω ότι η λειτουργία του κανονισμού αυτού, η εφαρμογή του κανονισμού αυτού θα πρέπει να εξασφαλίσετε και από χρηματοοικονομικής πλευράς. Ποιοι θα είναι λοιπόν οι πόροι που θα δοθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τα κράτη-μέλη προς την πρωτοβουλία αυτή, αυτό δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο και πρέπει αυτό να επισημαίνεται σαφώς στην γνωμοδότηση. Από την άλλη, πιστεύω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει η ε, σωστή εφαρμογή του κανονισμού αυτού, όχι απλώς η θεωρητική εφαρμογή του. Η Επιτροπή μας λοιπόν έχει γνωμοδοτήσει πολλά και στο παρελθόν και λέμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να λάβουν την κατάλληλη ενημέρωση για τον κανονισμό αυτό και ότι θα πρέπει να ενημερώνται για τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας που έχουν. Θα πρέπει να ληφθούν λοιπόν υπόψη οι γνωμοδοτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν από άλλους συναδέλφους της Επιτροπής μας ως προς αυτό. Θα πρέπει να γίνουν επίσης οι απαραίτητες αλλαγές όσον αφορά την χρηματοδότηση για την πρωτοβουλία αυτή, καθώς επίσης και την παροχή της απαραίτητης ενημέρωσης στους πολίτες. Ο επόμενος προπολογισμό θα πρέπει να προβλέπει και μια ξεχωριστή γραμμή, πιστεύω, προς αυτό. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα το οποίο μας απασχολεί είναι εν γέννη πολιτική επικοινωνίας και ενημέρωσης. Η Επιτροπή μας συζήτησε το ζήτημα αυτό πολύ συχνά, το συζητάει πολύ συχνά, όλες τις πιθανές πτυχές αυτές της πολιτικής επικοινωνίας, είτε πρόκειται για τις δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε πρόκειται για την διαφάνεια στην πολιτική επικοινωνίας. Ως προς λοιπόν αυτό το ζήτημα θα πρέπει να προβλέψουμε ότι δεν θα υπάρξει καμία δημοσιονομική περικοπή η ενημέρωση των πολιτών θα πρέπει να χρηματοδοτείται επαρκώς και στο μέλλον. Το τρίτο ζήτημα το οποίο μας απασχολεί και είναι σημαντικό για μας και το οποίο τονίζουμε και σε αυτή την γνωμοδότηση είναι η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Όλοι γνωρίζετε ότι αφοσιώσαμε πολύ χρόνο συζητώντας το ζήτημα αυτό στην Επιτροπή μας Αφιερώσαμε πολύ χρόνο, με συγχωρείτε. Αναφέρομαι εδώ στον κανονισμό για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων εν γέννη και σε ενδεχόμενες αλλαγές που θα προκύψουν στη χρηματοδότηση των κομμάτων αυτών στο μέλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να αναφερθεί στη γνωμοδότηση για το ζήτημα αυτό. Δεν γνωρίζω ακόμα τα τελικά αριθμητικά στοιχεία, πάντως ο προπολογισμός θα πρέπει να είναι έτσι ισορροπημένος, ώστε να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα χρήματα, απαραίτητη πόρη για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Η δική μας Επιτροπή πολλές φορές στο παρελθόν αναφέρθηκε στη σημασία του κανονισμού για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι πολύ σημαντική η χρηματοδότηση των κομμάτων αυτών για τη σωστή λειτουργία των ευρωπαϊκών ε, θεσμών. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίζεται για όλα τα ευρωπαϊκά, πολιτικά κόμματα ιδέουσα χρηματοδότηση. Θα συντάξουμε ένα ξεχωριστό κείμενο όσον αφορά ε, τις πηγές από όπου θα προέρχεται αυτή η χρηματοδότηση. Αυτά είναι τα σημαντικότερα σημεία της χρηματοδότησης αυτής. Η 4η Μαΐου είναι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 4 Απριλίου το μεσημέρι, στις 12 το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στις 23 και 24 Μαΐου για αυτή την γνωμοδότηση. Στη συνέχεια τον Ιούνιο και τον Ιούλιο θα έχουμε τη συνήθεια δικασία για τον προπολογισμό. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, διότι ο συνάδελφος Σαουντάργας είπε όλα τα θέματα που θεωρούμε και εμείς σημαντικά. Νομίζω ότι γενικά ζούμε σε ε, ένα καιρό που μπορούμε να βρούμε νέο χρήμα από αναδιατάξεις και όχι από νέα χρηματοδότηση. Και με την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών, με δικές μας πρωτοβουλίες μετά τη Λισαβόνα και με αυτά κυρίως που αποφασίσαμε για ε, το μελλοντικό καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, ξέρουμε ότι υπάρχει κόστος που συνδέεται με αυτό. Ε, κόστος βέβαια και ενημέρωσης αλλά και κόστος που υποστηρίζει την πραγματική πολιτική δουλειά για τους πολίτες που χρειάζονται ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να ενημερώνει τους πολίτες, να τους συμβουλεύει με υπηρεσία ιδιαίτερη, ξεχωριστή και μέχρι σήμερα ε, στο σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπεται το προσωπικό. Λοιπόν, χωρίς προσωπικό και χωρίς ε, υλικοτεχνική υποδομή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Περιμένω με ενδιαφέρον και ανυπομονησία τις προτάσεις και όλα τα υπόλοιπα τα συζητάμε όταν θα έχουμε το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Guerrero. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομος, διότι θεωρώ ότι το σχέδιο γνωμοδότησης διατηρεί την προσοχή στα θεμελιώδη ζητήματα που μας απασχόλησαν στην Επιτροπή ε, Συνταγματικών Υποθέσεων τους τελευταίους μήνες. Και θα πρέπει να δούμε και προς το μέλλον πώς θα κινηθούμε και πώς θα αναπτύξουμε νέες προτάσεις. Για άλλη μια φορά μιλούμε για ε, ανάγκη πραγματικής όμως επικοινωνίας με τους πολίτες και ε, την ανάγκη να υπάρχει και δημοσιονομική υποστήριξη γι' αυτό. Αυτό που ζούμε τους τελευταίους μήνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μας ε, επιβάλλει, μας συμβουλεύει να εξηγούμε στους πολίτες τι επιπτώσεις θα έχει για την καθημερινή του ζωή ε, αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που κάνουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θέματα συνταγματικά. Γνωρίζω ότι στο παρελθόν το θέμα αυτό γνώρισε την απόρριψη κάποιας ομάδας, αλλά ε, εξακολουθώ να πιστεύω και να επιμένω ότι η επικοινωνία αν είναι ειλικρινής, πραγματική και ουσιαστική είναι πάντα ένα στοιχείο σύνδεσης με τους πολίτες και με τη διαφάνεια ε, της λειτουργίας μας. Επίσης, η θέση σε ισχύ της πρωτοβουλίας πολιτών μας απασχόλησε πολύ στις εργασίες μας και όπως είπε μόλις ο, ο συντάξης νομοδότησης από πλευράς προϋπολογισμού θα πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, γιατί είναι κάτι που ε, εγκρίναμε πριν από λίγες εβδομάδες και αυτό είναι το νομικό καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ε, ό,τι έχει σχέση με τη χρηματοδότησή τους, κομμάτων και ιδρυμάτων. Ε, θα κάνω και καμιά τροπολογία, πάντως γενικά συμφωνώ με τον εισηγητή. Ο κύριος Ευχαριστώ. Θα ήθελα να φερθώ στο σημείο 2 του σχεδίου γνωμοδότησης που αναφέρεται στους πόρους για την επικοινωνιακή πολιτική υπέρ της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αναφέρεται εδώ πέρα όμως τίποτα κατά, δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το αρνητικό εδώ πέρα. Πιστεύω ότι πρέπει να αναφερόμαστε στα πραγματικά εδώ πέρα γεγονότα, ή μάλλον δίνεται η εντύπωση ότι να αφαιρεθούμε στα πραγματικά γεγονότα, θα αποφευχθούν πάρα πολλέ αρνητικέ εντυπώσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση που δήθεν οφείλονται στην άγνοια, ενώ στην πραγματικότητα οφείλονται πολλέ φορέ στη γνώση. Επίση, αναφερόμαστε σε περισσότερους πόρους που θα μπορούσαν να δοθούν για την επικοινωνική πολιτική, για άλλες υπηρεσίες, για άλλους φορείς. Δεν νομίζω όμως ότι ε, θα πρέπει να δοθούν πόροι για μια επικοινωνία η οποία ουσιαστικά θα είναι μια μονομερής προπαγάνδα όσον αφορά το σημείο 3 της γνωμοδότησης που αναφέρεται στη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Πιστεύω ότι σε έναν ιδανικό κόσμο τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τα μέλη τους και αυτό θα καταδεικνύει βασικά αν χαίρουν υποστήριξη ή όχι. Είμαι κατά της χρηματοδότηση των κομμάτων από διάφορες ενώσεις ή από επιχειρήσεις γιατί ουσιαστικά στη συνέχεια τα πολιτικά κόμματα πρέπει να ακολουθούν είναι τις επιταγές των επιχειρήσεων αυτών, των ενώσεων αυτών. Επίσης, η χρηματοδότηση πολλές φορές από τα ίδια τα κράτη κάνει τα πολιτικά κόμματα να ακολουθούν με ε, τρόπο πάρα πολύ πιστό τις επιταγές των κρατών αυτών. Βέβαια, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει χρηματοδότηση αυτή. Δεν θα πρέπει να, να είμαστε κατά της χρηματοδότησης αυτή στον ισχύ για κάποια κράτη-μέλη. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 4η Μαΐου το μεσημέρι για τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε κατά πάσα πιθανότητα στις 24 Μαΐου για τη γνωμοδότηση αυτή. Όσον αφορά τώρα την συνεδρίαση των συντονιστών σήμερα, δεν θα γίνει η συνεδρίαση αυτή γιατί ε, θα ξεκινήσουμε τη συνάντηση με τον κύριο Τρεμόντι σε 7 λεπτά. Δεν θα έχουμε τον χρόνο να συνεδριάσουμε. Χθε είχαμε μια πολύ σύντομη συνάντηση των συντονιστών. Ουσιαστικά συζητήσαμε την επίσκεψη της Επιτροπής μας στην Βαρσοβία, αναφερθήκαμε σε ποσοστώσεις. Ξέρετε, το Προεδρείο θα λάβει μια νέα απόφαση για το αν είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε την ποσόστοση που προβλέπεται. Περιμένουμε λοιπόν την απόφαση αυτή του Προεδρείου αν η απόφαση ληφθεί πριν την επίσκεψή μας, τότε θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την απόφασή μας. Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε είπαμε ότι ο κύριος Καζίνη θα πάει από το ΕΛΚ, Λεγκρίπ επίσης, από τους αλιστές Γκουρμάι Γκουρμάι-Ουγκερέρο και ο κύριος Ντάφα από τους Φιλελεύθερους και στη συνέχεια θα έχουμε τρία άτομα που θα έρθουν εκτός ποσοστώσεων ο κύριος Χέφνερ, ο κύριος Σόλτς και εγώ. Ελπίζω λοιπόν η διαφιλονικούμενη απόφαση του Προεδρείου να μην ληφθεί, γιατί η απόφαση αυτή δεν θα επιτρέπει επιπλέον άτομα να συμμετέχουν σε αυτή την επίσκεψη. Αυτά όσον αφορά την συνεδρίαση των συντονιστών, νομίζω ότι έχουμε ακόμα στη θέσή μας 6-7 λεπτά. Ας κάνουμε λοιπόν ένα σύντομο διάλειμμα, 6-7 λεπτά. Πιστρέψτε όμως παρακαλώ πολύ αμέσως μετά, γιατί ο κύριος Τρεμόντι θα ξεκινήσει την παρέμβασή του σε 11.30 ακριβώς. Να περάσουμε λοιπόν στο τελευταίο τμήμα της σημερινής συνεδρίασης. Είναι εδώ ο υπουργό Τζούλιο Τρεμόντι. Τον ευχαριστώ για την παρουσία του εδώ και τον χαιρετίζω εξ ονόματος όλων. Η συνάντηση αυτή ζητήθηκε από τον ίδιο τον Υπουργό και εγώ όταν μίλησα και με τους συντονιστές ε, των ομάδων. Ακούγομαι. Μήπω ακούγομαι καλύτερα με αυτό το μικρόφωνο. Ωραία. Χαιρετίζουμε λοιπόν τον Υπουργό, τον ευχαριστούμε για την παρουσία του εδώ. Το θέμα το οποίο θα ήθελε να θίξει αφορά ε, την Ευρώπη σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι αφορά τη σχέση μεταξύ της αλληλεγγύης ε, και της ε, πρακτικής της εφαρμογής και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αλληλεγγύη είναι η ψυχή της Ευρώπης, αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλληλεγγύη προς όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και η έννοια της αλληλεγγύης είναι γεγραμμένη σε δύο άρθρα της Συνθήκης της Λισαβόνας, το άρθρο 80 που αφορά εσωτερικές σχέσεις και το άρθρο 222 για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σοβαρή κρίση την οποία βιώνουμε, η οποία δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά όπως θα μας πει ο υπουργό αφορά και άλλους τομείς, ε, πλέον η παγκοσμιοποίηση αφορά και το Σύνταγμα και την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει έναν τρόπο για να εκφράσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ελληναγκή της, η οποία προβλέπεται στη συνθήκη της Λισαβόνα και αποτελούσε πάντα αναπόσπαστο τμήμα των καταβολών τη. Από τότε που οι ιδρυτές ε, σκέφτηκαν την έννοια τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Δεν θα ήθελα να καθυστερήσω άλλο αυτή τη συνάντηση. Ε, και γι' αυτό αμέσως μετά από την παρέμβαση του Υπουργού θα δώσω το λόγο για ερωτήσεις και παρατηρήσεις καταρχάς τους συντονιστές ε, της Επιτροπής μας ε, ή κάποιον εκπρόσωπο της κάθε πολιτικής ομάδας. Αν δεν μιλήσει ο συντονιστής θα μιλήσει κάποιο μέλος της πολιτικής ε, του ομάδας και αν υπάρχει χρόνος θα δώσουμε το λόγο στους υπολείπους. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας γιατί πρέπει να περατωθεί η συνεδρία στις 12.30 και εάν δεν υπάρχουν άλλοι αγορητές από τα μέλη της Επιτροπής θα, μπορούσαν να, θα μπορούσαν να παρέμβουν και άλλα μέλη. Ε, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς γιατί είναι τακτική συνεδρίαση αυτή. Σας δίνω το λόγο απευθείας κύριε Τρεμόντη. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Είναι τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα σε μια επιτροπή η οποία στην ονομασία της συνταγματικών υποθέσεων επισημαίνει το γεγονός ότι ε, υπάρχει ε, διαχωρισμός μεταξύ της συνταγματικής ε, συνθήκης και του συντάγματος. Και όλα αυτά, το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το όραμα των ιδρυτών της. Θα ήθελα σήμερα να μην ε, ακολουθήσω την πεπατημένη και να κάνουμε ένα τεστ αντοχής των συνθήκων και να σας εξηγήσω για ποιο λόγο θέλουμε να κάνουμε αυτό το τεστ αντοχής. Και θα σας ε, παραθέσω το Σέξπιρ εδώ. Υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα στον ουρανό και στη γη από όσα ε, διανοείται κανείς στη φιλοσοφία. Οι ευρωπαϊκές συνθήκες ενσωματώνουν το όραμα, το όραμα που, βρισκόμασταν, που είχαμε όταν βρισκόμασταν στην ηλικία της βεβαιότητας και τις γνώσεις. Η ζωή μας δίνει τη δυνατότητα να ζούμε όχι μόνο με βεβαιότητες και αστάθειες αλλά και, και σταθερότητα, συγγνώμη, αλλά και με αβεβαιότητα και αστάθεια. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να γίνει ένα τεστ αντοχής για να δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε το όραμα να σας πω εκ των προτέρων ότι εγώ θεωρώ ότι μπορούμε και θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε και θετικό αποτέλεσμα. Αλλά υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι η ερμηνεία και η εφαρμογή των συνθήκων θα πρέπει να γίνεται υπό το πνεύμα των καιρών που ζούμε. Υπό το πνεύμα της παρούσας κατάστασης και με το βλέμμα προς το μέλλον. Άλλωστε, για τα νομικά ζητήματα, στο νομικό τομέα, η ερμηνεία είναι ε, αέναη, εν εξελίξη. Η παρούσα ερμηνεία του ρωμαϊκού δικαίου είναι κατά πάσα πιθανότητα διαφορετική από την ερμηνεία που έδιναν οι Ρωμαίοι η ερμηνεία που δίνουμε εμείς σε ένα πίνακα του Ρέμπραντ είναι κατά πάσα πιθανότητα διαφορετική από την ερμηνεία που έδιναν οι σύγχρονοί του. Στους γάμους, όπως και στις συνθήκες, υπάρχει συνήθις δέσμευση ε, ότι κάποιος επισέρχεται στο γάμο και για τα καλά και για τα άσχημα. Καταρχάς να σας πω ότι ως προς τη μέθοδο στις συνθήκες ε, ασχολούμαστε ε, κυρίως με τα καλά στοιχεία. Η πρώτη ανάγνωση ενός συντάγματος μας δίνει μονίμως θετικά και καλά πράγματα. Ελευθερία, δημοκρατία, ελευθερία του ατόμου, ευημερία, βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική οικονομία της αγοράς, ε, τέλος στους διαχωρισμούς, παράλληλη πρόοδος προς το μέλλον. Η εντύπωση ότι στην πολιτική και νομική οικονομία των συνθήκων ε, δίνεται ότι πάντα το καλό είναι ο κανόνας και το κακό είναι η εξαίρεση. Στην πράξη όμως, στη ζωή έχουμε και το καλό και το κακό, και τη βεβαιότητα και την αβεβαιότητα. Υπάρχει πάντα ένα αρνητικό γεγονός. Ο τύπος του αρνητικού γεγονότος ε, στις συνθήκες περιλαμβάνεται σε ένα ε, κλασικό βασικό τύπο φυσικές καταστροφές ε, ή ανθρωπ... καταστροφές οι οποίες προκλήθηκαν από τον άνθρωπο. Από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες, πολιτικούς κινδύνους, ε, επιθώσεις, σειράξεις, ε, πολέμους, οικονομικές ανισορροπίες. Εάν το προσέξετε, πρόκειται για όρις οι οποίοι είναι οι ίδιοι από τα 1800 και είναι αναχρονιστικοί. Είναι πολύ συγκεκριμένη αυτή η περιπτωσιολογία και στην εξαίρεση του κακού δεν υπάρχει μια βαλβίδα ευελιξίας, δεν υπάρχει αυτό που οι Γερμανοί νομικοί αποκαλούν ε, το Μπεγκρίφ και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δώσουμε και εμείς μια ερμηνεία. Μια ερμηνεία η οποία πρέπει και μπορεί να είναι πολύ εκτεταμένη όπως γίνεται παραδοσιακά στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τρεις περιπτώσεις οι οποίες συσσωρεύτηκαν αυτά τα τελευταία δύο χρόνια και μας έφτασαν σε ένα ε, πολύ συχνό φαινόμενο, ε, πολιτικό φαινόμενο. Υπάρχει οικονομική κρίση, γεωπολιτική κρίση και η ατομική κρίση, πυρηνική κρίση. Κρίση, καταστροφή είναι ελληνικές λέξεις και από τα ελληνικά έρχεται και η βαθιά αίσθηση των αλλαγών. Η κρίση είναι αλλαγή του παραδείγματος και η καταστροφή είναι η αλλαγή της πραγματικότητας. να σας πω τώρα τα συμπεράσματά μου και να τα μοιραστώ μαζί σας. Στην οικονομική κρίση, στις συνθήκες, η νομική βάση είναι πολύ ευρεία, αλλά δεν είναι αρκετά ευρία. Η εφαρμογή που γίνεται για τη διαχείριση της κρίσης είναι πολύ ισχυρή. Στην περίπτωση της γεωπολιτικής κρίσης, το γράμμα της συνθήκης είναι πολύ ευρύ, αλλά η εφαρμογή της συνθήκης ε, στην πράξη θα μπορούσε να αποκληθεί και missing in action. Θα μπορούσε να, ε, ε, να το πούμε και με άλλο τρόπο. Missing in non-action. Δεν έχουμε δράσεις, δεν έχουμε πράξεις. Για την πυρηνική κρίση τώρα, μετά από την καταστροφή στη Φουκοσίμα, διαπιστώνουμε ότι τα όσα λέει η συνθήκη δεν επαρκούν και οι παρεμβάσεις, ακόμα και τα προληπτικά μέτρα, δεν μου φαίνεται ότι επαρκούν. Πιο συγκεκριμένα τώρα, για την οικονομική κρίση, Η οικονομική κρίση επί της αρχής έρχεται έξωθεν. Έχουμε τα όσα συνέβησαν στην παγκόσμια αγορά και μετά έχουμε οικονομικές συνέπειες στην Ευρώπη, χρηματοοικονομική κρίση κυρίως ε, στον ιδιωτικό τομέα. Εδώ λοιπόν είναι προφανές ότι στην Ευρώπη δεν υπήρχε ένα αποτελεσματικό κριτήριο μακροοικονομικής εποπτείας για τον ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό τομέα γινόταν έλεγχος των δημόσιων οικονομικών, ελλείμματα και χρέη, ε, γινόταν έλεγχος του πληθωρισμού, το καλάθι των αγορών, αλλά η αστάθεια που προκλήθηκε από τον ιδιωτικό τομέα δεν αποτελούσε αντικείμενο επαρκούς ελέγχου στην πορεία μου άκουγα συνέχεια όρους, υπερβολικό έλλειμμα, ε, πληθωρισμό στο καλάθι των αγορών, αλλά ποτέ δεν άκουσα για τη φούσκα το κτηματομεσητικού τομέα, τα πιστοτικές κάρτες ε, και πολλά άλλα. Η κρίση λοιπόν παρουσιάζεται και πρέπει με κάποιο τρόπο να τη διαχειριστούμε. Στις συνθήκες είναι πολύ συγκεκριμένη η ορολογία που χρησιμοποιείται. Μεγάλες διαταραχές στην οικονομική κατάσταση ενός κράτους μέλους, ε, μεγάλη επιδείνωση στην ε, προμήθεια συγκεκριμένων προϊόντων, και όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει δυσκολίες ή απειλείται από μεγάλες φυσικές καταστροφές ή εξαιρετικές περιστάσεις που είναι εκτός του ελέγχου του. Ποιος είναι ο χαλακτήρας αυτών των εξαιρέσεων. Οι εξαιρέσεις αναφέρονται όλες σε ένα κράτος μέλος. Είναι όλες περιπτώσεις κρίσης πριν από την ενιαία αγορά και ακόμα διαπιστώνουμε ότι έχουμε εξέταση αναχώρα. Δεν έχουμε γενικευμένη εξέταση της ανιάχωσης αγοράς. Αυτό που έγινε λοιπόν είναι να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε μια γενική προσέγγιση, να θεωρήσουμε ότι η κρίση ήταν ένα φαινόμενο το οποίο πλήττει όλα τα κράτη και όχι ένα μεμονωμένο κράτος. Δηλαδή θεωρήσαμε ότι έχει εξελικτική πορεία. Οι αλλαγές ήταν πολύ ισχυρές και κατά κάποιο τρόπο... Ε, ανεστάλλει το παράδειγμα της συνθήκης. Η συνθήκη της ε, Μάστρι, του Μάστρι, τη συνθήκη της Ρώμης και η διαχείριση της κρίσης ε, οδήγησε σε κορύφωση των χρεών και δημιουργήθηκε ένας μακρύς κατάλογος εξαιρέσεων των κανόνων. Δηλαδή και στη μακρό και στη μικροοικονομία η διαχείριση της κρίσης μας μετατόπισε από την οικονομία βάσης και μας δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα. Ας ελπίσουμε ότι ήταν αποτελεσματικό. Υπήρξαν ε, ευθύνε. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε τώρα. Η γεωπολιτική κρίση. Από τον Ατλαντικό στην Ασία άλλαξαν τα πράγματα. Αν θέλετε να είστε ενημερωμένοι, διαβάστε τη βίβλο το άνοιγμα των υδάτων. Η ένταση αυτών των ιστορικών γεγονότων, οι οποίες προκύπτουν από ένα ε, σύνολο παραγόντων και από την κερδοσκοπία ε, για τα τρόφιμα, αλλά υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες ε, δεν δέχονται τις απαγορεύσεις, οι νέοι που είναι πλέον ενημερωμένοι, η αντίδραση κατά κλεπτοκρατικών καθεστώτων, η ε, σχέση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλα αυτά δημιούργησαν μια λυσιδική αντίδραση γεγονότων και μια αλλαγή. Και αυτό φυσικά έχει και συνέπειες για τη δική μας Ήπειρο δεν περιορίζονται μόνο στο τμήμα που πάει από τον Ατλαντικό στον Αραβικό κόσμο και θα, φτάσει, και θα φτάσουν και στην Ασία. Και όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και στην Ήπειρό μας. Αν δούμε τα όσα λέει η συνθήκη και πάλι είναι πολύ ευρύ το λεξιλόγιο και καλύπτει σε μεγάλο βαθμό όλα αυτά. Βέβαια, πολλοί κανόνες έχουν εγγραφεί μετά από την 11η Σεπτεμβρίου για την τρομοκρατία, αλλά όλα πηγαίνουν προς την λογική της αλληλεγγύης. Η μεγάλη εισρωή ε, μεταναστών από τρίτες χώρες. Και εδώ δεν έχουμε μόνο το δικαίωμα στη μετανάστευση ενός ανθρώπου, έχουμε το συλλογικό φαινόμενο, το μαζικό φαινόμενο. Η συνθήκη επαρκεί όπως είναι γραμμένη. Η εφαρμογή της όμως μέχρι τούδε ήταν ανεπαρκή σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν μου φάνηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηλεφώνησε στις Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν νομίζω ότι το πολιτικό όραμα για τα θέματα αυτά είναι επαρκές. Είναι ανεπαρκές. Και δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων και επαναχρηματοδότησης, είναι πολύ πιο γενικό το ζήτημα στις τροχές του φόβου δημιουργούνται οι πολιτικές ισορροπίες της Υπήρου μας και αν δεν καταλάβουμε αυτή την αλλησυνειδωτή αντίδραση φαινομένων δυστυχώς ελοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε μια πολύ μεγάλη δημοκρατική αποδόμηση της, της Υπήρου μας. Και δεν νομίζω ότι το να αγνοήσουμε το φόβο των λαών και να θεωρήσουμε ότι είμαστε υπεράνω αυτών των αισθημάτων είναι ο σωστός τρόπος για να διαχειριστούμε δημοκρατικά αυτές τις πραγματικότητες. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ε, και να αφογκραστούμε τι νιώθουν οι λαοί αυτοί. Μπορεί να είναι και αβάσιμος ο φόβος τους, αλλά υπάρχει φόβος και θα πρέπει να έχουμε πολιτεία υπό την έννοια και της κατανόησης των αισθημάτων και των θελήσεων των λαών. Αλλιώς ε, είμαστε λανθασμένοι στις κρίσεις μας, είμαστε κοντόφθαλμοι. Γι' αυτό ακριβώ σα λέω ότι μέχρι τούδε η Ευρώπη ήταν missing in action. Παρά το γεγονός ότι στη συνθήκη υπάρχει μια ευρύτατη βάση δυνατοτήτων παρέμβασης. Εν τέλει, έχουμε την κρίση μετά από τη Φουκουσίμα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για ένα απλό τεχνικό ατύχημα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που έχει να κάνει με το Homer Simpson. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο ε, σημαντικό και έχει ιστορική βαρύτητα. βαρύτητα ε, είναι ένα γεγονός μακράς διάρκειας που δεν έχει σύνορα και που μας θέτει μεγάλα ερωτηματικά. Και επ' αυτού νομίζω ότι η συνθήκη δεν είναι καθόλου συγκεκριμένη. Αν δείτε το 20ο κεφάλαιο για το περιβάλλον, το 23ο κεφάλαιο για την προστασία των πολιτών, θα διαπιστώσετε ότι είναι ανεπαρκείς οι απαντήσεις που δίνονται. Γράφεται ο ρηπαίνων πληρώνει, η αρχή της πρόληψης, η αρχή ε, της ε, προσοχής, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να υλοποιούνται και να μην μείνουν κενό γράμμα. Είμαστε βέβαιοι ότι συμβαίνει αυτό. Είδαμε τι γίνεται με τα πυρηνικά. Έχουν καταγραφεί για μας ε, ε, τα στοιχεία αυτά. Έχει καταγραφεί το κόστος για τις συντάξεις μας σε 50 χρόνια. Το κόστος του παροπλισμού έχει καταγραφεί. Έχουμε υπολογίσει το ασφαλιστικό κόστος. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, τοπικά προβλήματα, αλλά ε, τα δεινά είναι παγκόσμια και θα πρέπει ε, να γίνει μια εξέταση για τα πυρηνικά θέματα. Μπορούμε άλλωστε να το κάνουμε. Υπάρχει κάτι για τα πυρηνικά, αλλά δεν υπάρχει στη συνθήκη της Ρώμης. Υπάρχει στη συνθήκη Βρατών που νομίζω ότι είναι ακόμα ακόμα Και εκεί υπάρχει το δικαίωμα των κρατών να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες, να ζητήσουμε έρευνες, να εφαρμόσουμε τα κριτήρια της πρόληψης. Και νομίζω ότι όλα αυτά είναι θεμελιώδη. Για να είμαι πιο σαφής, Νομίζω ότι αν κάνουμε τον απολογισμό ε, για όλο το κόστος και για όλα όσα μπορούμε να κάνουμε είναι ε, η κατάλληλη χρονική στιγμή να το κάνουμε, η ιστορική στιγμή. Έχουμε το παλιό διαβόητο σχέδιο, να έχουμε ε, σχέδια και επενδύσεις για την έρευνα και την καινοτομία και να γίνει και η διάσημη μελέτη για τη Μεσόγειο και να χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά τα προγράμματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με ευρωομόλογα. Νομίζω όμως ότι μακρηγόρησα για να επανέλθω στις συνθήκες. Μία έκκληση σας κάνω. Μην σταθούμε μόνο στη διαλεκτική στο Χέγγελ μεταξύ ισχύω και έλλειψης ισχύω, ας ε, δούμε την κοσμοπολιτική θεωρία του είναι και την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Νομίζω ότι καλύπτεται ένα μακρύ φάσμα και νομίζω ότι μας δίνεται και μια νέα ερμηνεία, ε, ένα αμάλγαμα προβλημάτων τα οποία συνδέονται και τα οποία επιτρέπουν, ε, μας ζητούν να ζητήσουμε περισσότερη Ευρώπη και όχι λιγότερη Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν η Ευρώπη η οποία θα πρέπει να σκεφτεί εις βάθος αυτά τα προβλήματα, να ταρκουνηθεί, να ξεκινήσει εξ αρχής και να σκεφτεί τον εαυτό της χωρίς εθνικούς εγωισμούς αλλά ταυτόχρονα και τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, ε με εξέπληξε ιδιαίτερα αυτός ο συλλογισμός σας που λέει ότι θα πρέπει ε, να προάγουμε τις χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή πλήττονται από την ε, ε, ένδια και το φόβο και ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να τις σκεφτούμε. Αν κατάλαβα καλά αυτό που είπατε, να δώσω το λόγο αμέσως γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας σε όσους ζήτησαν να μιλήσουν. Καταρχάς λοιπόν, εξ του ΕΛΚ, ο κύριος Μπρόκ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για τις εκτενέστατες ε, παρατηρήσεις και την παρουσίαση ότι το ευρωπαϊκό όραμα πρέπει να αντέξει στις ε, δοκιμές αντοχής και στο στρες και να αποδείξει την ύπαρξή του. Αλλάζουν οι καιροί και θα πρέπει να αποδείξει την ύπαρξή της Ευρώπη και είπατε ότι ε, απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν αρκεί το έθνος κράτος να το πράττει μόνο του, μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε από την ιδέα αποδυνάμωσης των κρατών για να μην μπορούν να ξανακάνουν πόλεμο. Αλλά τώρα έχει αλλάξει η κατάσταση. Θα πρέπει να είμαστε από κοινού σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις τρομοκρατίας, ενεργειακής ασφάλειας, μετανάστευσης, κλιματικής αλλαγής κλπ. Και στις διάφορες συζητήσεις που γίνονται, το είπατε στο τέλος, στα κράτη μας, θα πρέπει να συζητήσουμε τα πάντα μετά την καταστροφή στην Ιαπωνία, ας πούμε, συζητάμε την εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας. Αλλά θα πρέπει να δούμε αυτό τι συνέπειες θα έχει και σε άλλους τομείς. Μπορούμε να έχουμε ενεργειακό ε, ανεφοδιασμό σε προσιτές τιμές και εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες του κόσμου ολόκληρου. Αν έρθουν οι αναπτυσσόμενες χώρες ε, στο δικό μας επίπεδο θα τετραπλασιαστεί ανάγκη και κατανάλωση ενέργειας. Η μετανάστευση καταλαβαίνουμε ότι έχει αλλάξει. Ο κόσμος δεν έχει πια προοπτική ανάπτυξη στη χώρα του, ε, είτε είναι αυτό στη Βόρεια Αφρική, είτε είναι γενικά στην Αφρική. Και σε ε, καταστάσεις κλιματικής αλλαγής. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σημαίνει ε, ότι αυτό θα ε, φέρει σε αντιπαράθεση την ενεργειακή πολιτική με την πολιτική καλλιέργειας φυτών για τρόφιμα ή μήπως θα καταστρέψουμε τα παρθένα δάση. Ε, όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και να καταλήξουμε σε μια συνολική ανάλυση και του κόστους αλλά και του κινδύνου και όχι με μονομένα παραδείγματα. Αυτό οδηγεί και σε κάτι άλλο, σωστά το είπατε, ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους λαούς εδώ Και αν θέλετε να δούμε και το θέμα της μετανάστευσης, ε, πρέπει να δούμε και κάποιο ορισμό και να καθορίσουμε όταν είναι κλασικοί ε, πρόσφυγες που έχουν δικαίωμα ασύλου, καλώς. Όταν κινδυνεύουν γιατί διώκονται για πολιτικούς, ε, φιλετικούς, θρησκευτικού οποιουσδήποτε λόγους. Έχουμε πρόσφυγες που φεύγουν από τη χώρα τους γιατί θέλουν να γλιτώσουν από τον πόλεμο. Αλλά έχουμε και οικονομικούς πρόσφυγες, οικονομικούς μετανάστες. Σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την επιβάρηση της Ιταλίας δεν ξεκαθαρίζεται αυτή η διαφορά. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι οι μετανάστες από την Τινησία δεν είναι ούτε άτομα που αιτούν άσυλο, συγγνώμη, ε, ούτε πρόσφυγες. Ο σκοπός είναι να γυρίσουν πίσω στην Τινησία κάποια στιγμή, όχι να τους μοιράσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δείτε, γιατί υπάρχει μια σύγχυση και την επιβάρηση των μεμονωμένων κρατών. Στη δεκαετία του 90, στον πόλεμο των Βαλκανίων, η χώρα μου επί δύο-τρία χρόνια, κάθε χρόνο δεχόταν 800.000 πρόσφυγες. Ε, και δεν ένιωσαν καθόλου ευρωπαϊκή ελεγγύη το 2010 στη Γερμανία κατέθεσαν άσυλο 47.000, στη χώρα σας νομίζω 8.000, έτσι το 10. Και αυτό νομίζω ε, δεν συζητείται, γίνονται διαφορετικές συζητήσεις από χώρα σε χώρα, αλλά και αυτό βοηθάει για την εξέβρεση αλήθειας και θα πρέπει να βρούμε μια συνεννόηση συνολική για να καταλάβουμε πώς επιβαρύνονται οι μεμονωμένες χώρες και πώς θα εξισωθεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Όχι όμως με αποσιώπηση των αριθμών, δεν μας βοηθάει αυτό, γιατί ο καθένας θα πρέπει να το εξηγήσει και στη χώρα του και αν δεν μπορεί να το εξηγήσει θα έχει προβλήματα και ίσως να το λάβουμε και αυτό υπόψη στη συνολικότερη ανάλυση. Ευχαριστώ πολύ. E Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπροκ. Ο κύριος Γκουαλτιέρη στη συνέχεια, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ εξ ονόματος της ομάδας μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Τρεμόντι για την παρέμβασή του και διότι θέλησε να παρουσιάσει ανάλογες σκέψεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο θεσμικό όργανο το οποίο δεσμεύεται περισσότερο από όλου ε, στην προσπάθεια να μεταφράσει τις αρχές της αλληλεγγύης που είναι εγγεγραμμένες στη συνθήκη σε συγκεκριμένες δράσεις μέσω της ε, συνήθους νομοθετικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το γεγονός ότι παρενέβη εδώ ενώπιον της Επιτροπής Ταγματικών Υποθέσεων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η συνθήκη της Λισαβόνας έχει ως επίκεντρο, όπως υπενθύμησε και ο πρόεδρος Καζίνη, την αλληλεγγύη. Το άρθρο 83, το άρθρο 4.3, ε, αλληλεγγύη προς τα κράτη-μέλη, αλληλεγγύη ως αρχή βάση της οποίας θα πρέπει να υπάρχει μια πραγματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η αλληλεγγύη μεταφράζεται πιο συγκεκριμένα μέσω της σωστής ερμηνείας και σε αυτό συμφωνώ. Σωστή ερμηνεία των συνθήκων, συνθήκε οι οποίε μα επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε συνήθι αλλά και ε, πιο ασυνήθιστα μέσα για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Και εδώ είμαστε υπέρ τη πρώτη άγουσα που είναι η άγουσα που ακολουθούμε μέσω τη κοινοτική μεθόδου. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στου τρει ε, τομεί στου οποίου αναφέρθηκε ο Υπουργό. Όσον αφορά την οικονομική διάσταση, είμαστε αυτή τη στιγμή εντός μια πολύ δύσκολη συζήτηση για την υιοθέτηση του πακέτου της διακυβέρνησης και του governance και εμείς εδώ στην Επιτροπή μας προσπαθήσαμε να αποφύγουμε το πέρασμα από την νομική βάση του άρθρου 122.2 για την αλληλεγγύη προβλημάτων του δημοσίου χρέους και υπάρχει ένα νέο άρθρο της συνθήκης στα κράτη-μέλη το οποίο επιτρέπει ένα μηχανισμό σταθερότητας και αυτό δεν θα είχε συμβεί χωρίς την κοινοτική μέθοδο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να, υπάρχει, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει αλληλεγγύη μέσω της κοινοτική μεθόδου. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο θέμα, εδώ έχουμε δύο δρόμους. Το άρθρο 80, το οποίο επιτρέπει και μάλιστα επιβάλλει να χρησιμοποιηθεί το στοιχείο της αλληλεγγύης στην εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων, τη διαχείριση του ασύλου, τη διαχείριση των πολιτικών μετανάστευσης. Και εδώ νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολύ λίγα για να προετοιμαστούμε, για να αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης από τα κράτη-μέλη με ε, το, την Ιταλική κυβέρνηση εξ αρχής που θα έπρεπε ούτως ή άλλως να είχε κατευθύνει αυτή τη συζήτηση στο Συμβούλιο και να φτάσουμε μέχρι και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου έχει καθήκον όχι πέραν του ε, δικαιώματος νομοθετικών προτάσεων τις οποίες θα πρέπει να υλοποιήσει και να χρησιμοποιήσει για τον τομέα αυτά. Υπάρχει επίσης και το άρθρο 22 το οποίο και αυτό με τη σειρά του επειδή ακριβώς ε, αφορά αφορά έκτακτα φαινόμενα ζητά μια πιο διακυβερνητική αντιμετώπιση η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ακραία περίπτωση παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιείται και σε αυτές τις περιπτώσεις αλλά περιλαμβάνει και μια πιο συνηθισμένη ε, πτυχή και λέει στην τελευταία παράγραφα ότι το Συμβούλιο αξιολογεί τακτικά τις απειλές τι οποίες θα μπορούσε να δεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λοιπόν ελπίζουμε το Συμβούλιο να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη διάταξη του Συμβουλίου και επομένως να κάνει τακτική αξιολόγηση των δυνητικών απειλών. Και τέλο, όσον αφορά το τρίτο στοιχείο, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά για τι ισχύουσε συνθήκε, ξεκινώντα από διαφορετική αντιμετώπιση από πλευρά Συμβουλίου όσον αφορά την ε, μελλοντική διάσταση του ευρωπαϊκού προπολογισμού, χωρί ε, τον οποίο η δέσμευση αυτή ε, η οποία εκφράζεται από πλευρά Υπουργού για τις επενδύσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δύσκολα θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι καθόλου διατεθειμένο να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση, όπως άλλωστε και κάνει, και ελπίζουμε η παρέμβαση αυτή του Υπουργού να μεταφραστεί και σε δράση από πλευράς Ιταλικής κυβέρνησης στο Συμβούλιο και μια καλύτερη στάση του Συμβουλίου επί των θεμάτων αυτών. Θα ήθελα επίσης από τον Υπουργό να είναι λίγο πιο συγκεκριμένος, διότι στην παρέμβασή του αναφέρθηκε και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις της συνθήκης οι οποίες ε, ίσως να είναι απαραίτητες, αλλά οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν και υπό το συγκεκριμένο πρίσμα ε, του να υπάρχει ομοφωνία που είναι πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή ως έχει κατάσταση. Θα πρέπει κυρίως λοιπόν να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή της ισχύουσας συνθήκης. Ευχαριστώ τον κύριο Καλτιέρη και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ντάφ ε, εξ ονόματος των Φιλελευθέρων. Oh, Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα τον κύριο Τρεμόντι γιατί αποφάσισε να έρθει εδώ και να μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός χώρος για να παίρνει κανείς το λόγο και για να γίνονται τέτοιες συζητήσεις για τα θεμελιώδη αυτά ζητήματα. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει ως ένα, μια ομοσπονδιακή στιγμή που πρέπει τελικά να αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε ακολουθώντας τον ομοσπονδιακό δρόμο ή αν θα οπισθοδρομήσουμε, αν θα επιστρέψουμε σε πιο εθνικι, εθνικές, εθνικιστικές τάσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό ζήτημα το οποίο τίθεται σε όλα τα κράτη-μέλη και εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό εδώ στις Βρυξέλλες. Η ελληνική πάνω απ' όλα απαιτεί αμοιβαία εμπιστοσύνη. Και θεωρώ ότι υπάρχει μία απουσία ισχυρής αμοιβαία εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή. Γενικά, οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τις συνθήκες της Λισαβόνας και νομίζω τελικά δεν εμπιστεύονται οι μεν τους δε. Επομένως διανύουμε μια πολύ σημαντική κρίση. Και η κρίση αυτή φαίνεται πάρα πολύ στα πλαίσια της εγχώρησης της εσωτερικής πολιτικής των κρατών μελών, όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, διάφορα εθνικά πολιτικά κόμματα, τα οποία δεν καταφέρνουν πλέον κατά την άποψή μου να υποστηρίξουν την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με τρόπο δημοκρατικό και με τρόπο αποτελεσματικό. Στο τέλος της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της υφιστάμενης τρέχουσας της θητείας, θα πρέπει να είμαστε σε θέση, πιστεύω, να έχουμε προχωρήσει σε ένα πακέτο μεταρρυθμιστικών μέτρων όσον αφορά το Σύνταγμα, συνταγματικών μέτρων. μέτρα τα οποία θα πρέπει να δυναμώσουν τον πυλώνα της οικονομικής διακυβέρνησης, μέτρα τα οποία θα πρέπει να δημιουργήσουν μια κοινή αγορά για, την, για τον ενεργειακό εφοδιασμό, μέτρα τα οποία προσπαθήσαμε να συζητήσουμε και στα πλαίσια πραγματεύσεων για τη συνθήκη τη Λισαβόνα, χωρίς όμως θετικό αποτέλεσμα. Και πιστεύω, και αυτό το είπε και ο κύριος Γουαλτιέρη, ότι θα απαιτηθεί τελικά μία πιο ευέλικτη μέθοδος προκειμένου να προβαίνουμε στο μέλλον σε στεγματικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί του παρόντος έχουμε παραλύσει από το γεγονός ότι ε, οποιαδήποτε αναθεώρηση της συνθήκης θα πρέπει να χαίρει τη σύμφωνη γνώμης και της επικύρωσης όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίσαμε τι προβλήματα προκάλεσε αυτό για τη συνθήκη της Λισαβόνας και είμαι πεισμένος ότι αν δεν κάνουμε κάτι προκειμένου να καταστήσουμε το σύστημα λίγο πιο ευέλικτο, τότε θα συναντήσουμε το πρόβλημα αυτό εκ νέου στο μέλλον. Θα ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων λοιπόν αν καταφέρναμε τελικά να είχαμε εκ μέρους της Ιταλικής κυβέρνησης μία σαφή συμβολή ως προς αυτό, προκειμένου να εμβαθύνουμε λίγο τη συζήτηση όσον αφορά τις ε, τροποποιήσεις που μπορούμε να επιφέρουμε στο μέλλον στη συνθήκη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντάφ. Ο κύριος Χέφνερ τώρα για τους Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Υπουργό Τρεμόντι για την παρουσία του εδώ σήμερα. Και ε, πέρα από τα θέματα της επικαιρότητα και της καθημερινότητας μας εξηγήσατε και γενικότερα πώς βλέπετε την Ευρώπη και οραματικά. Μ' αρέσει αυτό. Δεν θα πρέπει να αντιδρούμε με βάση επίκαιρες κρίσεις ή καταστάσεις, έτσι να σερνόμαστε πίσω από τις εξελίξεις, αλλά να βλέπουμε πώς θέλουμε να διαμορφώνουμε και το μέλλον. Θα ήθελα να σημειώσω τρία θέματα από όσα αναφέρετε. Το πρώτο, εσείς επεκταθήκατε πολύ το θέμα του μηχανισμού διάσωσης, του μηχανισμού ε, σταθερότητας και την οικονομική διακυβέρνηση και την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών και στην Ευρώπη, αλλά κατ' επέκταση και τι γίνεται με το ευρώ. Αν σας κατάλαβα καλά, θα ήθελα να υπογραμμίσω και τη δική σας αίσθηση ότι η κρίση δεν είναι ουσιαστικά στον πυρήνα της μια κρίση του δημοσίου τομέα αλλά στην Ευρώπη έχουμε πλέον αναπτύξει μια σταθή κατάσταση που επεκτείνεται συνεχώς και συμπεριλαμβάνει και άλλους τομείς και θα ήθελα να σας διαβιβάσω και τις ανησυχίες μου. Για ποιο λόγο αγωνιώ εγώ. Παίρνουμε μέτρα, σταθεροποιούμε το επίγον, αλλά δεν έχουμε φτάσει σε εκείνο το στρώμα βάθους που είναι η ρίζα του κακού. Δηλαδή, επιβαρύνουμε και πάλι το δημόσιο τις δημόσιες υπηρεσίες, τις υποδομές, τις κρατικές επενδύσεις στο μέλλον. Ε, ε τις περιορίζουμε ακριβώς επειδή έχουμε επιβαρύνει το δημόσιο τομέα. Και από την άλλη τα κέρδη ιδιωτικοποιούνται και μάλιστα καλπάζουν τα ιδιωτικά κέρδη. Αυτό δεν είναι κακό, δεν είναι σφάλμα, αλλά είναι ανισορροπία. Το ίδιο ισχύει με την εξέλιξη του εισοδήματος στα κράτη-μέλη μας. Είναι όλο και δυσκολότερο να ζει κανένας από τον ιδρώτα του προσώπου του, για να το πω έτσι, από τη δουλειά του, για τη χειρονακτική. Στα χαμηλά στρώματα ε, χαμηλώνει το εισόδημα και ε, σε κάποιους άλλους αυξάνεται, οι οποίοι δεν εργάζονται, απλώς επενδύουν και τοποθετούν τα χρήματά τους και στη συνέχεια εμείς δανείζουμε χρήματα στις τράπεζες ακριβώς για να τις σταθεροποιήσουμε αλλά ε, αποδυναμώνεται και η πολιτική και ο δημόσιος τομέας όλο και περισσότερο ενώ αυξάνουν ε, οι τόκοι συνεχώς ε, και υπάρχει μια μετατόπιση, μια νέα διανομή του πλούτου προς τους ιδιώτες. Αυτό με μένα με ανησυχεί, με τρομάζει. Θα πρέπει λοιπόν πέρα από τα έκτακτα μέτρα να σκεφτούμε και τι επιπτώσεις έχουν αυτά τα μέτρα που παίρνουμε για να σώσουμε μια κατάσταση, για να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιστρέψουμε με άλλο τρόπο ε, που να έχει νόημα και κοινωνικό αλλά και σε θέματα ελευθερίας, ίση πρόσβαση, ε, ευκαιρίες, δικαιοσύνη, δημοκρατία. Μια κατεύθυνση που να είναι πιο ε, παραδεκτή και πιο αποδεκτή, να στρέψουμε προς εκεί τις εξελίξεις, γιατί φοβάμαι ότι θα χάσουμε όλο και περισσότερο τη στήριξη των πολιτών μας. Και πιστεύω κι εγώ, όπως και ο Άντρου Ντάφ, αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Και έγινε μία πρόταση και για τη Λισαβόνα, για μελλοντική μέθοδο, μια συντακτική συνέλευση, γιατί τώρα μπαίνουμε σε μια νέα φάση ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι μέσα χρειαζόμαστε, τι εργαλεία, αλλά στο κάτω-κάτω και τι Ευρώπη θέλουμε, προς τα πού θέλουμε να στραφεί η Ευρώπη, σε ποια κατεύθυνση και πώς μπορούν να το κάνουν τα θεσμικά όργανα και οι μηχανισμοί τους οποίους ε, υιοθετούμε. Και πολύ σύντομα, έχω δύο ακόμα. Το ένα είναι η Φουκοσίμα, η πυρηνική ενέργεια, σωστά είπατε ότι και το κόστος που προκαλεί ο παροπλισμός, η εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας είναι σημαντικό. Αλλά θα ήθελα να πω ότι είναι τεράστιο το κόστος της μη εγκατάλειψης πυρηνικής ενέργειας και να το συμπληρώσω με μία σκέψη έτσι, αρχής. Στην πολιτική των δημοσίων οικονομικών, όπως και εδώ, ακολουθούμε μια ε, πολιτική μετά από μένα το χάος μετά από μένα ο κατακλυσμό και για περίμηχθή το. Να βγάλω εγώ τώρα όσα μπορώ και άλλο να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Ναι, αλλά το κόστο που μεταθέτουμε στο μέλο με τόσα τεράστια ποσά, ποσότητα συγγνώμη, αποβλήτων που ε, προσπαθούμε να αποθηκεύσουμε, να το παρακολουθούμε, αυτό είναι ένα βάρος που μεταθέτουμε σε επόμενες γενιές και πολλές γενιές. Και αυτό θα το βρούμε ε, μπροστά μας. Είναι μια επιβάρυνση των επομένων γενεών. Εμείς έχουμε ε, χρέος να παραδώσουμε ένα πλανήτη καθαρό, βιώσιμο στις επόμενες γενιές. Και οικολογικά στέκει μόνο να χτίζονται, να κατασκευάζονται νέε πυρηνικέ μονάδε, νέα πυρηνικά εργοστάσια, μόνο εφόσον υπάρχει μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία που να ασφαλίζει 100% ε, του κινδύνου για οποιοδήποτε ατύχημα. Και απορώ πως δεν έχει γίνει μέχρι τώρα κάτι τέτοιο. Αλλιώς, όχι, στα πυρηνικά. Τώρα, έχουμε επιστήμονες των οποίων οι απόψει δίστανται, αλλά θα πρέπει να ακούμε και τι δύο πλευρέ. Να ακούμε και του επιστήμονε εκείνου που στέκονται πιο επικριτικά απέναντι στην πυρηνική ενέργεια, για να ενισχύουμε την εμπιστοσύνη εκεί που τη χάσαμε να την ανακτήσουμε στι πολιτικέ αποφάσει. Το τελευταίο θα το αφήσω, γιατί δεν έχω χρόνο για να μιλήσουν και οι συνάδελφοι για να απαντήσουν. Αλλά ήθελα να αφαιρθώ σε αυτό που είπε ο Μπροκ, το θέμα τη αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά του πρόσφυγε. Είμαι πολύ υπέρ της αλληλεγγύης, αλλά μην είναι μέτρο ad hoc, επίγον και έκτακτο. Να σκεφτούμε η Ευρώπη πώς ε, δεν θα γίνει ένα ανάλγητο φρούριο, αλλά μια ανοιχτή ένωση ε, και συνέπειες ε, της ευημερία μας να επεκτείνονται και γεωγραφικά. αλλιώ είναι δραματικές οι εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ. Μας πιέζει ο χρόνος και θα πρέπει νομίζω να κάνω αυτό που σας είχα πει στην αρχή. Δηλαδή θα δώσω το λόγο μόνο στα μέλη της Επιτροπής μας. Έχω τρεις ακόμα ομιλητές, αλλά είναι όλες από την ίδια πολιτική ομάδα. Α, συγγνώμη, να δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Σόλτς και μετά τον κύριο Μοργκάντη. Έχουμε λοιπόν μόνο έναν από τους συντηρητικού και δημοκράτες από, τους, ε, συγγνώμη, από την ομάδα της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Να ζητήσω συγγνώμη από τους κυρίους Πιτέλα και Αντζελίλη, ε, δεν, δεν μπορώ να σας δώσω το λόγο, δεν σας χαιρέτησα και στην αρχή, συγγνώμη, σας χαιρετώ τώρα. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να σας δώσω το λόγο γιατί πρέπει ακόμα να, ακούσουμε, να ακούσουμε τον κύριο Σόλτς και τον κύριο Μοργκάντη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και σας Υπουργέ ευρύτατη συζήτηση γίνεται για όλα τα θέματα που μας ε, προβληματίζουν και μας απασχολούν καθημερινά. Και θα πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον της Ευρώπης να έχουμε μια ε, ειλικρινή και ισότιμη μεταχείριση και των επόμενων γενεών θα πρέπει να το συζητάμε σε μεγαλύτερο βάθος και πιο συχνά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια όταν συζητούμε ευρωπαϊκά ζητήματα. ακριβώς αυτούς τους καιρούς που επικρατεί μεγάλη ανασφάλεια στον πληθυσμό. Αν δείτε τα τελευταία αποτελέσματα των εκλογών σε κάποια κράτη-μέλη φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι δεν θεωρούν ότι τους εκπροσωπούν οι παραδοσιακές ε, απαντήσεις του πολιτικού κόσμου και των πολιτικών ε, ελίτ εν γέννη και του συστήματος. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι θέλει η πολιτική, τι πράττει η πολιτική, γι' αυτό τελικά το χάσμα μεταξύ των πολιτών ε, και της πολιτικής διευρύνεται συνεχώς. Και αυτό φτάνει μέχρι και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλήσατε για το Σπινέλη, ένα από τους ιδρυτές ε, πατέρες της ευρωπαϊκής κοινότητας τότε και οραματιζόταν με τη συνθήκη της Ρώμης να επέλθει η ειρήνη για τους λαούς της Ευρώπης και η συνύπαρξη, η συμβίωση ουσιαστική και προσπάθησε να βάλει και μια προοπτική για τη δικαιοσύνη και για τις επόμενες γενναίες. Ακριβώς σήμερα καλούμαστε αυτό το όραμα και ε, αυτή την εντολή και το καθήκον που μας μεταβίβασε ε, ο Σπινέλη να το κάνουμε πραγματικότητα. Κατά πόσο τα έργα μας συνάδουν με τα λόγια μας. Μιλάμε απλώς για τη συνεργασία στην Ευρώπη ή την εφαρμόζουμε κιόλα. Θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας όχι μόνο την πολιτική αλλά και τους εταίρους μας, τους συνομιλητές μας, τους πολίτες και τις προσδοκίες και τα όνειρά τους. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον συνάδελφο Άντρου Ντάφ που λέει ότι ήδη από τώρα ε, η επομένη ε, ημέρα μια συνθήκη είναι η προηγούμενη ημέρα της επόμενης ίσως. Θα πρέπει να σκεφτούμε δηλαδή ε, πώς θα αντιμετωπίζουμε τέτοια θέματα ε, κρίση, διάσωση τραπεζών, οικολογικές προκλήσεις, πυρηνική ενέργεια. Πώς θα φτάσουμε στην αηφορία, στην αηφόρο χρήση της ενέργειας και πώς θα πείσουμε και τον κόσμο να είναι στο πλευρό μας. Και να αναφέρω και κάτι που δεν υπόθηκε ακόμα Είμαι πεπισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ευκαιρία ε, να ε, υπάρξει μόνο αν είναι κοινωνική Ευρώπη. Αν έχουν δηλαδή εμπιστοσύνη οι πολίτες για την καθημερινότητά τους, επαναλαμβάνω, ότι μπορούν να ζουν από την εργασία τους, να τραφούν, ε, να ζήσει η οικογένειά τους και να έχουν ευκαιρία και τα παιδιά τους και οι νέες γενιές σε όλα τα κράτη-μέλη. Με όραμα, με προοπτική και για το μέλλον να μπορούν να ζουν οι άνθρωποι. η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει πραγματική ουσιαστική οικονομική ένωση και καθημερινή ή θα είναι μια νομισματική ένωση και εν μέρη οικονομική. Πώς θα έχουμε μια οικονομική πολιτική και κοινωνική πολιτική που θα συνδέει το εθνικό με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Γιώσκα Καφίσερ μίλησε στη Λέσχη Σπινέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπε ότι όταν μιλάμε για την Ευρώπη θα πρέπει να σκεφτόμαστε τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, μιλήσατε κι εσείς για το όραμα που είχαν οι ιδρυτές πατέρες. Δεν ξέρω χρειαζόμαστε Ηνωμένε Πολιτείε Ευρώπης. Δεν είμαι εγώ αυτός. Αλλά εμείς θα πρέπει να απαντήσουμε στο εξή ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τούτη εδώ, έχει το σθένος και τη δυνατότητα να αναπτύξει μια πολιτική που να είναι ε, μια πολιτική κοινωνικής δικαιοσύνης με κοινωνικής Ισότητα, ε, κοινωνική ισότητα. Ελλάδα, ε, Πορτογαλία, Ιρλανδία, ε, Σονία. Και μια τελευταία παρατήρηση για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε συνέπεια στην πολιτική αλλά και συνέπεια μεταξύ των διαφόρων τομέων και πεδίων της πολιτικής και μια ειλικρίνεια στη συμπεριφορά μας και στη σχέση των τριών θεσμικών οργάνων με βάση την ισχύουσα συνθήκη. Και έχω την αίσθηση ότι το Συμβούλιο δεν έχει καταλάβει, έχει τεθεί σε ισχύ το Συμβούλιο, το, η συνθήκη συγγνώμη της Λισαβόνας, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως άμεσα εκλεγμένος εκπρόσωπος του λαού έχει λόγο για ορισμένες ε, κοινοτικοποιημένες ε, πολιτικές και έτσι αυξάνεται και η δημοκρατική νομιμότητα. Και αυτό είναι ένα θέμα αλληλεγγύης και πάλι μπορεί να συζητηθεί η σχέση της κοινοτικής μεθόδου με την διακρατική. Αυτό πρέπει να το λύσουμε αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που είναι παγκόσμιες αλλά και ευρωπαϊκές. Κυρίως πάντα υπέρ των πολιτών. Ευχαριστώ κύριε Σόλτς και τέλος ο λόγος στον κύριο Μοργκάντη. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, καταρχάς καλωσορίσατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξ ονόματος ε, της Ομάδας Ελευθερίας της Δημοκρατίας. Έχουμε μεγάλη αύξηση στα ποσοστά των ε, ευρωσκεπτικιστών κομμάτων. Ακούσαμε το μεγάλο ποσοστό που πήρε το Φιλανδικό Κόμμα των Ευρωσκεπτικιστών που θα μπορούσε να τον οδηγήσει και στην κυβέρνηση της χώρας του. Σε ένα από τα σημεία λοιπόν του προγράμματος του Πολιτικού Κόμματος των Φιλανδών ήταν η χρηματοδότηση ε, για τη διάσωση χωρών όπως η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Τι γνώμη έχετε εσείς για αυτό το μέτρο, πώς θα μπορούσε να διασωθεί η Ευρώπη και πιστεύετε ότι υπάρχουν ε, ε, δυνητικοί κίνδυνοι καταρχάς για το ευρώ και κατά δεύτερον για την ε, όλη πολιτική και οικονομική και νομισματική σταθερότητα της Ευρώπης. Τελευταία ερώτηση. Θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει μέτρα διαχωρισμού μεταξύ των ε, τραπεζών ε, που κάνουν συναλλαγές και των ε, τραπεζών αποταμιευτηρίων, όπως για παράδειγμα τα όσα συνέβησαν στην αντίστοιχη Αμερικανική Τράπεζα. Να δώσω τώρα το, το λόγο στον Υπουργό για να απαντήσει. Εγώ δεν έχω να θα σας θέσω κάποια ερωτήματα, εκτό από μια ερώτηση ουσία, ε, όμω, την οποία δεν μπορώ να κρατηθώ και θα σα την κάνω. Τον τελευταίο καιρό ο τύπο αναφέρθηκε στη θέση τη Ιταλία, η οποία είναι ε, μια θέση ευρωσκεπτικιστική. Δηλαδή, ε, υπήρξαν κάποιες ε, δηλώσεις και αναφέρθηκε και η ιδέα της ε, εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω την εντύπωση, κύριε Υπουργέ, ότι η δική σας η τοποθέτηση είναι τελείως διαφορετική. Είναι η τοποθέτηση ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει την Ιταλία ως ιδρυτικό μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατανοεί ότι είναι τεράστια τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά θεωρεί ότι είναι μια ευκαιρία για να δώσουμε μια νέα όθηση στην Ευρώπη, η οποία απαιτεί φυσικά και κόπο αλλά και ψυχή. Και να υπενθυμίσω και την συζήτηση που έγινε μετά από την πτώση του τείχους του Βερολίνου και ακούστηκε ότι είδαμε ένα μηχανισμό με τέλειους ε, τροχούς αλλά δεν μπόρεσα να βρω πουθενά την ψυχή και η αλληλεγγύη αποτελεί τμήμα αυτής της ψυχής. Δεν ξέρω αν κατανόηση την έννοια της παρέμβασής σας αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι το περιεχόμενο των όσων μας είπατε. Ο Υπουργός, ευχαριστώ. Άκουσα έξι παρεμβάσεις, όλες πολύ ενδιαφέρουσες. Ε, η πρώτη παρέμβαση ήταν του κυρίου Μπροκ. Νομίζω ότι την πρώτη παρέμβαση λοιπόν του κυρίου Μπροκ η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ακούστηκε μία πολύ σο σωστή θέση για τη μέθοδο. Ακούσαμε όλα τα υπέρ και τα κατά ε, για όλα τα ε, όσα βιώνουμε και όσα εκδηλώνονται και αυτά είναι σωστά. Θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς έχει το κόστος, πώς έχει ε, η εναλλακτική λύση και τι πλεονεκτήματα υπάρχουν όταν επιλεχθεί η εναλλακτική λύση. Είναι πολύ νωρί για να κάνουμε απολογισμό, αλλά είναι αρκετά νωρί για να αρχίσουμε να κάνουμε την ανάλυση του κόστους, του θετικού κόστους και των θετικών στοιχείων. Πρόκειται για φαινόμενα τα οποία συνέβησαν όλα εν μία νυχτή. Μέσα σε τρία χρόνια έχουμε τρει πολύ έντονε αλλαγέ. Yes. Και αυτό λοιπόν είναι σωστό αυτό που μας προτείνεται. Να κάνουμε ε, μία ε, ισορροπημένη ανάλυση. Να σα πω κάτι για να είναι σαφέ. Εγώ δεν έχω έρθει εδώ για να ζητήσω χρήματα για τους μετανάστε. Κάνω μία εντελώ διαφορετική συζήτηση. Εγώ θα ήθελα να επαναληφθεί η ιστορία με τις τέλειες ταυτότητες. Να επα... Θα ήθελα τα όσα συνέβησαν στα Βαλκάνια να είναι συγκρίσιμο με όσα συνέβησαν στη Μεσόγεια. Πρόκειται όμως για φαινόμενα τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερα ιστορική ένταση. Δεν είναι επεισοδια... Ε, φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν για δύο χρόνια έχουν πολύ σημαντική ιστορική βαρύτητα και θα πρέπει να τα εξετάσουμε και υπό αυτό το πρίσμα. Ο κύριος Γκουαλτιέρη θέτει το ζήτημα του κατά πόσον ε, θα πρέπει να ξεφύγουμε από τις συνθήκες για να δημιουργήσουμε μια νέα συνθήκη. Και αυτό το ερώτημα τίθεται και από τον κύριο Νταφ νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε ως ενδεχόμενο. Θα ήθελα να είμαι πολύ σαφής. Οι συνθήκες γράφτηκαν πριν από την παγκοσμιοποίηση. Προσαρμόστηκαν περιθωριακά, αλλά είναι προϊόν ενός παρελθόντος κόσμου τότε ο κόσμος αποτελούνταν από το ευρωπαϊκό μπλοκ, από το σοβιετικό μπλοκ, από το αμερικανικό μπλοκ. Σε κάποιες συνθήκες νομίζω δεν αναφερόμαστε πολύ συγκεκριμένα στην Ασία και στην Ανατολή. Ο κόσμος έχει αλλάξει εκ βάθρων. Ίσως η κρίση η οποία δημιουργεί ασυνέχεια λόγω αλλαγής παραδείγματος μπορεί να μας οδηγήσει σε μία νέα και πιο έντονη συνθήκη. Να δράξουμε την ευκαιρία λοιπόν. Ο κύριος Χέφνερ θέτει ένα ζήτημα το οποίο ξεκινά από την οικονομία Είναι αρκετά διαφοροποιημένη η διαχείριση που, ε, που έγινε. Έχω την τύχη να μιλώ ε, από πλευράς μιας χώρας που δεν χρειάστηκε να κάνει ε, μια αλλαγή λόγω της κρίσης. Εμείς όμως πέραν κάποιων ε, κοινωνικών παρεμβάσεων δεν χρειάστηκε να κάνουμε δημόσιες διαπάνες για να διαχειριστούμε την, κρίση παρά το γεγονό ότι υπήρξαν προβλήματα. Σε άλλες χώρες ε, χρειάστηκε να γίνουν παρεμβάσει. Στο New Deal του Roosevelt ε, σώσαμε τις επιχειρήσεις, τους ιδιώτες και ε, τις οικογένειες. Σε αυτή τη διαχείριση της κρίσης διασώσαμε τις τράπεζες εις βάρος των οικογενειών. Είπαμε ότι οι τράπεζες είναι δομικό στοιχείο και γι' αυτό κάναμε τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για το μετά. Εγώ θεωρώ ότι εμείς στην Ευρώπη θα πρέπει να αναλογιστούμε λίγο πώς έχει το οικονομικό μας μοντέλο και επομένως και το κοινωνικό μας μοντέλο. Μπορεί να είναι ένα μοντέλο το οποίο θα διέπεται αποκλειστικά από τη ζήτηση για καταναλωτικά αγαθά μπορεί να είναι ένα μοντέλο το οποίο θα διέπεται αποκλειστικά από τις εξαγωγές. Δεν νομίζω. Θεωρώ ότι ένα τραπέζι για να στέκεται όρθιο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία πόδια και αυτό θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και για δημόσιες επενδύσεις που χρηματοδοτούν δημόσια ζήτηση για συλλογικά αγαθά. Και οι παρεμβάσεις για τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αυτής της μορφής οι παρεμβάσεις που αναζητούμε κοινωνική οικονομία της αγοράς. Αυτό έχει σημασία. Αναφερόμαστε στην οικονομία της αγοράς χωρίς την κοινωνική πτυχή, μόνο όταν αναφερόμαστε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν ξέρω γιατί χάθηκε το κοινωνικό στοιχείο εδώ, αλλά στη συνθήκη αναφερόμαστε στην κοινωνική οικονομία της αγοράς. Και νομίζω ότι αυτή είναι η ισορροπία μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών της Υπήρου μας. η οικονομία καθορίζεται ως προς το στυλ της για τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός ε, προέκυψε από ένα ε, ε, Ιταλό που είναι ο οικονομικός λογαριασμός αφενός και ο κληρονομικός λογαριασμός. Το οικονομικό είναι το τι θα ξοδέψουμε σε μια χρονιά και το κληρονομικό είναι το τι θα αφήσουμε ως κληροδότημα στις μελλοντικές γενναίες. Επομένως θα πρέπει να βασιστούμε και στις δύο πτυχές. Να μην σκεφτούμε μόνο την οικονομική πτυχή και τους λογαριασμούς, αλλά να σκεφτούμε και το τι θα αφήσουμε ως κληρονομιά. Για να μην αφήσουμε κινδύνους μόνο στις μελλοντικέ γενναίες, αλλά και θετικά στοιχεία. Ο κύριος Σόλτς έθεσε το ερώτημα τις σχέσεις μεταξύ της ιδέας που έχουμε για την Ευρώπη ως λαοί και του τι σχέση έχει αυτό με την κρίση. Εγώ είμαι αρκετά μεγάλο και θυμάμαι αυτέ τι παλιέ ταινίε που μα έδιναν μια δυναία τη Ευρώπη. Βλέπουμε τι Ιψίκαμίνου τη Γεωργία, ε, το γάλα που ήταν προϊόν ε, ενός ε, κόσμου ίσω παρελθοντικού αλλά ξέρετε όλοι ότι το γάλα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο θερμό από το επιτόκιο. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε και κάποια στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με την εργασία, με τη χειρονεκτική εργασία και όχι μόνο με τα οικονομικά και τα χρηματοπιστωτικά. Ο κύριος Μοργκάντη έκανε μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Είναι στην επικαιρότητα η υποβάθμιση και η αρνητική ε, βαθμολογία των οικονομικών των ΗΠΑ. Και όχι μόνο οι ειδήσει που έχουμε για τις εκλογικέ αναμετρήσεις, που είναι εξίσου σημαντικές, αλλά είναι σημαντικέ και αυτές οι ειδήσει. Θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν και τα αίτια των ψήφων αυτών προς τέτοια κόμματα και τα αίτια τα οποία μας οδηγούν σε ανάγκη για πιο ευρύ ασφάλιση. Η άποψή μου είναι ότι αν λύσουμε, εάν μπορούμε να λύσουμε θέματα για περιφερειακές χώρες, από εκεί και πέρα το μπλοκ της Ευρώπης θα μπορέσει να ε, εκφράσει τα όσα θέλει μέσω ευρωπαϊκών ομολόγων. Για τους ευρωσκεπτικιστές τώρα, είπατε ότι ε, κάποια πράγματα για την άνοδό τους συμφωνώ με την άποψή σας. Ο Πρόεδρος, νομίζω ότι ήταν πολύ επικοδημητικά τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι έδωσαν τροφή για σκέψη σε όλους εμάς από την Επιτροπή. Ευχαριστώ όλους. Πέρα στη συνεδρία.